Αμέσως. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα αφού συναντηθήκαμε χθε ξανά για τη συζήτησή μας και σε ομάδες εργασίας και, στην αυριανή, και στη βραδινή συνάντησή μας συναντηθήκαμε Θερμό καλωσόρισμα στον Πρωθυπουργό τον κύριο Ορμπάν που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόσο. Έχουμε επιφανείς καλεσμένους και βασικούς ομιλητές σήμερα στην διακοινοβουλευτική αυτή συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πρόεδροι, είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας σε αυτή την κοινοβουλευτική μας ε, συνάντηση και το θέμα είναι τα Δυτικά Βαλκάνια προς μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη. Πολύ σημαντικό θέμα για όλα τα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Έγινε πολύ καλή συζήτηση χτες. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα έχουμε 21 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις επίσημες γλώσσες και κροατικά, βοσνιακά, σερβικά, μακεδονικά, αλβανικά κλπ. Και μπορείτε ε, να συμπληρώσετε τα έντυπα για χρόνο αγόρευσης αν θέλετε αγαπητοί συνάδελφοι να πάρετε το λόγο στη συζήτηση. θα υπάρξει συζήτηση ε, με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας και προεδρία του Συμβουλίου τον κύριο Όρμπαν και με τον κύριο Μανουέλ Μπαρόσο, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά λοιπόν τώρα στην αρχή της συνεδρίασής μας και θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο τον κύριο Κέμπερ επειδή είμαστε συμπρόεδροι βλέπετε στη συνεδρίαση ε, να πάρει, να μιλήσει. Ευχαριστώ Λάσλο που ήσουν πάντα αποτελεσματικός και συνεργάσιμος εκ μέρους της Ουγγρικής Προεδρίας και σου δίνω λοιπόν την Προεδρία της συνεδρίασης. Ε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Τιμή για μένα αυτή και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε όλοι στη δεύτερη μέρα τη Συνόδου μας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το ανέφερε ήδη, χτες είχαμε πολιτιστική εκδήλωση και το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι εκθέσεις των ομάδων εργασίας που θα αναφέρονται στις χθεσινές εργασίες. Κάθε ομάδα εργασίας θα έχει ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή της για να παρουσιάσει αυτά που έκανε. Καταρχάς να ζητήσω από την κυρία Ντόρις Πακ να μας κάνει μια παρουσίαση των εργασιών της πρώτης ομάδας εργασίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε των διαφόρων θεσμικών οργάνων, αγαπητοί συναδελφοί, χθε είχαμε την ομάδα εργασίας 1 που ασχολήθηκε με τη συνεργασία στον τομέα του χώρου της ε, ελευθερίας, ε, δικαιοσύνης ε, και δημοκρατίας. Και τα θέματα της μετανάστευσης, ε, συνεργασίας αστυνομικών ε, υπηρεσιών κτλ. Κόπα και Πιεσκόφσκα είχαν συμμετάσχει και τόνισαν τη σημασία μεταξύ της, ε, τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας για τον τομέα της ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Δέκα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα μέλος από την Ανατολική Ευρώπη είχαν συμμετάσχει στη συζήτηση για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί μετά από τις εκλογές εκεί κοινοβούλιο και δυστυχώς δεν μπορώ να κατανοήσω το πώς ε, δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν και μόνο από πλευρά της Σερβίας και πάλι θέλω εδώ να πω η Πολωνία η Ουγγαρία, το Πέδιο, σχολίασαν τα θέματα της απελευθέρωσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ένα σημαντικό βήμα για την περιφερειακή συνεργασία και το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου ανέφερε τις προσπάθειες που γίνονται εκεί για να βελτιωθεί η ικανότητα να μπορέσουν να ενταχθούν στον οδικό χάρτη road map μετανάστευση, θέματα ασύλου ήταν διαρκώς θέματα κοινή συζήτησης. Η Γερμανία και η Ελλάδα εξέφρασαν ιδιαίτερα θέσεις όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο. Σε σχέση με τη συνάρτηση με το άσυλο και την παράνομη μετανάστευση, επίσης υπενθυμήθηκε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι σεβαστές αρχές η νέα πολιτική που καθορίζεται και με τη συνθήκες της Λισαβόνας θα πρέπει για το άσυλο να μπορέσει να λειτουργήσει πράγμα το οποίο ανέφεραν η Βουλγαρία και η Πολωνία. Επίσης αναφέρθηκε από πολλούς ότι η απελευθέρωση από διαβατήριων ε, δεν είχε σαν αποτέλεσμα να περάσουν πολλοί μετανάστες στις βόρειες και άλλες χώρες χάρη στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Από πλευράς Frontex έγινε θετική αξιολόγηση από τη Σουηδία, Ελλάδα και Ουγγαρία. Αστυνομική συνεργασία. Συνεργασία αστυνομική και συνεργασία περιφερειακή είχε σημαντικό ρόλο συζητήσεις. Η Πολωνία ήθελε περισσότερες λειτουργικές δυνατότητες συνεργασίας με τις χώρες αυτές. Μέχρι τώρα και για την Κροατία υπάρχει ε, κάποια ε, δυνατότητα εμπλοκής και αποστολές οι αστυνομικέ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Υπογραμμίστηκε το πολύ σημαντικό έργο σε σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε άλλους τομείς στα θέματα περιφερειακής συνεργασίας, Τα θέματα καταπολέμησης διαφθορά και της καταπολέμησης του εμπορίου ανθρώπων είναι προτεραιότητα στην αστυνομική συνεργασία για τη Σουηδία η πηγή όλων των κακών βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν λειτουργεί σε μια χώρα μια κοινωνική τάξη πραγμάτων σωστή όταν η οικονομία δεν βαίνει καλώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα κοινωνική τάξη πραγμάτων και κοινωνική ασφάλεια θα ήταν σημαντικά θέματα για την πρόληψη αυτό υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα από την Τσεχία η Σουηδία ιδιαίτερα είχε επιμείνει στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της σημασίας της Ευρωπόλ είναι κοινή συνένεση ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρέπει να ελέγχουν την υλοποίηση της εφαρμογής των νομικών αρχών για τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο ε, εργαστήριό μας, στο σεμινάριό μας. Και σε σχέση και με την Βουλγαρία και το σχόλιο που έγινε για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων επίση Δικαστικό σύστημα. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο είναι προτεραιότητα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα δικαστικά όργανα είναι κύριε ανησυχίε και μελήματα για όλους. Η εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαρκού εποπτείας για να ελέγχεται η συμμόρφωση με τι διατάξει Και η Βουλγαρία και η Ουγγαρία ζήτησαν να υπάρξει ένα τέτοιο μηχανισμό εποπτείας από από την άλλη πλευρά η συνεργασία με τη Σερβία σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία είναι κέρια σημασίας και αυτό σε σχέση με τα θέματα που ε, καλούνται εκεί και εξετάζονται εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Όλα θα πρέπει να ε, μπορούν να λειτουργήσουν και να συγκλίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν εύκολο. Αυτό ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πακ και τώρα θα στραφώ προς τον κύριο Μιχαήλ Μπάλα να μας πει τι έκανε η δεύτερη ομάδα εργασίας για την ένταξη των πολιτών αυτών των θέματων εργασιών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχα την τιμή να προεδρεύσω και να δώσω έκθεση για την ένταξη σε σχέση με τις εργασίες της ομάδας, ε, την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας εργασίας 2. Για τους Ούγγρους γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε μια ιστορία που μας δίδαξε ότι το να είναι κανείς πολίτης δεν είναι μια νομική ιδιότητα, αλλά εμπλέκεται κανείς συναισθηματικά, υπαρξιακά έχει και μια πολιτιστική διάσταση και ε, αυτή μεταξελίσσεται και είναι σημαντικό αυτό για την διαδικασία διεύρυνσης. Οι πολιτικοί πρέπει να γεφυροποιούν, να γεφυρώνουν να είναι γέφυρες ώστε οι νομικές αυτές κατηγορίες σε σχέση με τους πολίτες να προσεγγίζουν κάθε μέρα περισσότερο τους πολίτες. Για την Ουγγαρία είναι πιο εύκολο αυτό για μας γιατί έχουμε ιστορικούς δεσμούς ε, με τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε αναπτύξει ένα είδος αμοιβαία κατανόησης μεταξύ μας και γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα ως το θέμα της ε, κοινή κοινοβουλευτικής μας αυτής συνεδρίασης από πλευράς ε, Κάτσιν ε, Ευρωβουλευτό που ήταν συμπρόεδρος ε, τονίστηκε ότι η ολοκλήρωση και ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων έχει κέρια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι μια κύρια πρόσθετη αξία για την Ευρώπη που θα απορρεύσει συνολικά. Στις αρχικές τους παρεμβάσεις μας υπενθύμησαν την πολιτισμική πολυμορφία της πρώην Ιουγκοσλαβίας και τις χώρες που την συναποτελούσαν επιστήθηκε η προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις και κάποιος κατακαιρματισμός ακόμα που μπορούμε ακόμα να ε, ψηλαφίσουμε και να διαπιστώσουμε ότι υφίσταται σε αυτή την περιοχή, σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες από κοινού μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο συζητήσεις δεν θα βοηθήσουν με κανένα τρόπο να προαρθεί η αμοιβαία κατανόηση και συνεννόηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πολυμερές πλαίσιο, ένα φόρμα, ένα βήμα πολυμερές όπου πολυσχηδώς θα μπορούν να παρεμβαίνουν όλοι. Για να υπάρξει μια εξισορροπημένη παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες από πλευρά τη. Τονίστηκε επίση ότι τα διεθνή και θεσμικά όργανα και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πολλέ φορέ πόρο απέχουν από τα άτομα, από του πολίτε. Και σε σχέση με, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, αυτά τα κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για να, είναι, να γεφυροποιούν τι διαφορέ και να προσεγγίζουν του πολίτε περισσότερο. Στην εναρκτήρια παρέμβασή μου ανέφερα, αναφέρθηκα στην πρόοδο των Δυτικών Βαλκανίων. Υπό το πρίσμα του σε ποιο βαθμό αυτές οι χώρες συμμορφώθηκαν με οικονομικά, ε, νομικά, κοινωνικά κριτήρια. Για μια επιτυχή όμως ολοκλήρωση χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα. Την ένταξη και ολοκλήρωση όλων των πολιτών πλήρως και αυτό πρέπει να προχωρήσει και σε σχέση και με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Εξετάζοντας την ιστορία των τελευταίων 100 ετών στα Δυτικά Βαλκάνια, αυτό που μπορεί να δει κανείς είναι ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή την περιοχή. Μείωση δηλαδή των σειράξεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ εθνοτικών ομάδων. Γι' αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η ολοκλήρωση είναι η μόνη εναλλακτική λύση που απομένει στις χώρες αυτής της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Διότι η κοινωνία θα μπορέσει έτσι να δεχθεί τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ε, γνωρίζοντας ότι η ολοκλήρωση θα σημαίνει αμοιβαία κατανόηση, πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι εγκατάληψη της ταυτότητάς τους. Και το ίδιο ισχύει και αν, αν, αντίστροφα. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Η προσέγγιση και η κατανόηση των πολιτών θα είναι κάτι θετικό σε σχέση με την αποδοχή του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει να καταβάλουμε προσπάθειες να ευδοκιμήσει αυτός ο στόχος. Αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά η εκπαίδευση, η παιδεία είναι το πιο συνετό, το πιο σκόπιμο μέσο για να χρησιμοποιηθεί ώστε να υπάρξει πρόσβαση και να αλλάξουν πολλά πράγματα στο μέλλον. Φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ευκαιρία. Βλέπουμε ότι μεγάλη, ε, μεγάλος αριθμός μαθητών των Δυτικών Βαλκανίων θα ήθελε να δραχθεί της ευκαιρίας, θα επιθυμούσε να, να σπουδάσει στην ε, Ευρώπη. Φυσικά υπάρχει οικονομική δυσπραγία και τα κονδύλια δεν επαρκούν. Πρέπει να υποστηρίξουμε όμως αυτή την προσπάθεια, να τονωθεί αυτή η συνιστόσα. Ίσως θα πρέπει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από πλευράς κυβερνήσεων να προετοιμαστούν έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να γνωρίσουν καλύτερα οι νέοι τους πολιτισμούς των άλλων χωρών. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό θα σημαίνει ε, ότι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ε, ε, απουσίας ή αποχώρησης των νέων από αυτές τις χώρες. Χρειάζονται δίκτυα, διαδικτύωση. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να γυρίζουν στις πατρίδες τους και όχι να φεύγουν από αυτές και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους εκεί. Η πολιτισμική πολυμορφία πρέπει και αυτή να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί και αυτό είναι κύρια προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εκπρόσωποι των εθνοτικών ομάδων στα Δυτικά Βαλκάνια Βαλκάνια στην ευρύτερη περιοχή θα βλέπουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σαν μια οδό προ την ειρήνη. Είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η ελπίδα για τους πολίτες αυτής της περιοχής ότι δεν θέλει να συγχωνεύσει και να ισοπεδώσει αυτές τις παραδόσεις και πολιτισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμενη την πολυμορφία του πολιτισμικά θέλει να εντάξει αυτή της ε, παραδόσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, και σε σχέση και με την κληρονομιά, την φυσική κληρονομιά και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένα είδος εμπλουτισμού. Κάνουμε λόγο για την ένταξη και ολοκλήρωση με τους πολίτες. Στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι δεν, είναι, δεν πρόκειται μόνο για θέματα πολιτών μιας χώρας. Κάνουμε λόγο και για εθνοτικές μειονότητες ή εθνοτικές ομάδες εθνοτικές ομάδες και μειονότητες που ζουν και στις δύο πλευρές ε, ε, συνόρων, συνοριακών γραμμών, μεθοριακών γραμμών. Και αυτό πρέπει πάλι να λαμβάνεται υπόψη, ότι βρίσκονται μειονότητες ένθεν και ένθεν. Και είναι κέρια σημασία αυτό, να διασφαλιστεί αυτή η πολυμορφία. Όχι εις βάρος, όχι ως απειλή, αλλά ως ευκαιρία. Ως ευκαιρία της οποίας πρέπει να δραχθούμε υπήρχαν αντιπαραθέσεις σε σχέση με αυτές τις ομάδες και τριβές μεταξύ τους. Για τους κατοίκους όμως αυτής της περιοχής είναι κάτι το φυσικό και φυσιολογικό ότι πολιτισμοί και γλώσσες και παραδόσεις πρέπει και μπορούν να ζουν δίπλα-δίπλα η μία ε, δίπλα στην άλλη. Και έτσι από πλευράς μας είχαμε συνεισφορές από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που παρενέβησαν στη συζήτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να εμπλακούμε διάλογο με τις χώρες αυτής της περιοχής, συζητώντας τις πολιτισμικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που έχουν σημασία ιδιαίτερη για να υπάρξει προώθηση, προαγωγή της κατανόησης μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Το θέμα της εκπαίδευσης και της παιδείας τονίστηκε. Το να φροντίσουμε και να μεριμνήσουμε για τους νέους είναι κλειδί για την επιτυχία στο μέλλον. Αναφέρθηκε επίσης ότι συνταγμένες προσπάθειες θα πρέπει να προαθούν ώστε να προωθηθεί η κατανόηση, αλληλοκατανόηση μεταξύ των εθνοτικών ομάδων. Η πολιτισμική πολυμορφία πρέπει στα μαθήματα, στα ίδια τα σχολεία να προαθεί, ώστε να γαλουχηθεί η νέα γενεά, να είναι πιο ανεκτική, να δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι αυτοί οι νέοι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και παρακολούθησης συνοδευτικά μετά την, την αποχώρησή τους από το σχολείο. Είναι θλιβερό αλλά υπάρχει πάρα πολύ ψηλό ποσοστό ανέργων νέων σε αυτή την περιοχή. Φυσικά και η κατάσταση των φτωχότερων πολιτών πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό είναι ευκταίο μια πολιτική για τους Τσιγκάνους, τους Ρωμά, υπό την Ουγγρική Προεδρία να μπορεί να καλύπτει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων επίσης. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική για τη λεκάνη του Δούναβη θα πρέπει να μπορεί να προαγάγει αυτές τις πτυχές πολύμορφα. Όχι μόνο επιλύοντας και αντιμετωπίζοντας πολιτισμικά θέματα, αλλά παρέχοντας και ένα πρόγραμμα πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει και θα εντάσσει πολλά θέματα. Ο πολιτισμός ε, βλέπουμε είναι οι πολιτισμικές παραδόσεις ε, η πιο σημαντική δύναμη σε αυτή την ολοκλήρωση. Γι' αυτό είναι θλιβερό το ότι αυτή η πτυχή δεν την χάνει πάντα επαρκούς προσοχής σε σχέση με άλλες πολιτικές που ε, καλλιεργούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από τους συμμετέχοντες υπεγράμισαν θέματα λογοτεχνίας, μουσικής, ζωγραφικής, καλών τεχνών, οικαστικών, σημαντική πτυχή και αυτή της αμοιβέ κατανόησης. Διότι εργαζόμαστε υπέρ της ειρήνης. Για την ειρήνη από κοινού. Είναι σημαντική ευθύνη αυτή για όλους μας. Αν δεν μπορούμε να εντάξουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιληθούν αυτές οι σειράξεις και να αντιμετωπιστούν αυτές οι τριβές. Κάποια προσωπικά βιώματα, προσωπικές εμπειρίες αναφέρθηκαν σε σχέση σχέση με αυτή την περιοχή, τονίζοντας πάντα τη σημασία της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων. Αξίες, ταυτότητα, αρχές και αξίες και η ταυτότητα είναι τα κύρια στοιχεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να σα πω κάτι τεχνικό χαρακτήρα, λέει ο Πρόεδρο. Την εξή παρατήρηση. Ότι η μετάφραση από τα βουλγαρικά δεν είναι στο 21 αλλά είναι στο 17 διάβλος 17 για να ακούτε μετάφραση στα βουλγαρικά και τώρα θα πρέπει να καλωσορίσουμε με όλη μας την καρδιά τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας τον κύριο Όρμπαν ο οποίος θα μας ε, μιλήσει από πλευρά της κυκλικά εναλλασσομένης Προεδρίας Ένωσης Örülök annak, hogy egy, az Európai Unió bővítése είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το να μιλώ από αυτή τη θέση ε, σε εσά εδώ. Ε, είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην διεύρυνση. Η Ουγγρική Προεδρία και αυτή επομένω ακολουθεί την ίδια γραμμή πλεύση. Οπότε θα ήθελα τώρα, αν μου επιτρέπετε, να σα ε, αναφέρω τα εξή. Πρώτα-πρώτα, να δούμε ποιο είναι το όραμα που έχουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το όραμά μας είναι το εξής. Να είμαστε ρεαλιστές. Η αφετηρία μας είναι πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα. Μιλούμε για έναν θύλακα. Έναν θύλακα στην Επαϊκή Ήπειρο. Μιλούμε για μια περιοχή η οποία γειτονιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον ΝΑΤΟ, χώρες του ΝΑΤΟ και της Ένωσης. Μιλούμε για μια περιφέρεια όπου ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε. Και όταν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαμε για επανένωση της Ευρώπης, ενοποίησή της. Ο κομμουνισμός και ο Σόβιετ μεξάλαστ. Μιλούμε για μια διαδρομή που ξεκίνησε το 1945, μια τραγωδία, ε, ο κομμουνισμός, η Σοβιτική Ένωση και όλα αυτά διορθώθηκαν. Επρόκειτο για ένα προτσές που κανείς δεν αμφισβήτησε. Προσπαθούσαμε να ξαναβρούμε την πολιτιστική μας ενότητα. Να συνενώσουμε αυτά τα οποία επέπρωτο να είναι μαζί. Τώρα όμως Μιλούμε για μεγαλύτερες διαφοροποίησεις. Μιλούμε για διαφορές που είναι βαθύτερες. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν οι χώρες της Δύσης. Είναι τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα. Πάντως πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις μας. Θέλουμε πραγματικά τα Δυτικά Βαλκάνια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί ότι αυτό έχει κρυθεί. Ότι αυτό κρίθηκε τότε που Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές για μας ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια Ευρώπη με μαύρες τρύπες. Όλα αυτά υπονομεύουν την ασφάλεια, την ενότητα. Και εάν δεν σπεύσει η Ευρώπη να ενοποιήσει, θα σπεύσουν άλλοι. Ένα άλλο ζήτημα τώρα είναι κατά πόσον έχουμε σωστό χρονισμό. Εάν έχουμε σωστό timing για αυτά τα διαβήματα. Τι θα να κάνει η Ευρώπη, να διευρυνθεί ή να εμβαθύνει. Βλέπουμε ότι η σκακέρα αναδιατάσσεται συνέχεια παντού στον κόσμο όσον αφορά την ισορροπία των δυναμίων. Επομένω και εμεί να μην ξεχνούμε ότι οι προκλήσει είναι πάρα πολύ μεγάλε στην παγκόσμια σκηνή, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα πρέπει να κάτσουμε και να εξετάσουμε τι μπορεί να κάνει την Ευρώπη πιο ισχυρή. Η εμβάθυνση ή η διεύρυνση. Υπάρχει εμπειρία σε αυτό το επίπεδο γιατί όταν έγινε η διεύρυνση προς Ανατολάς τότε διαπιστώθηκε ότι το θέμα δεν είναι ή να κάνουμε το ένα ή να κάνουμε το άλλο αλλά πρέπει να κάνουμε και τα δύο και η διαδικασία της εμβάθυνσης και η διαδικασία της διεύρυνσης η μία ενισχύει την άλλη επομένως διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται να έχουμε ανανέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Άρα επομένως βλέπουμε τι γίνεται με ε, τις διαφορετικά, τα διαφορετικά εθνικά δίκαια, βλέπουμε τις διαφορετικές περιπτώσεις όπως θα υποβληθούν προς εξέταση σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ε, πάντως, θα πρέπει να δούμε πώς η διεύρυνση θα μας φέρει και καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Κάτι άλλο τώρα το οποίο ανάγεται στην εμπειρία μας, ανάγεται στην πρόσφατη διεύρυνση, είναι οι διαπραγματεύσεις για 21 και 1 και πλέον κεφάλαια. Θυμάμαι ήμουν εγώ τότε πρωθυπουργό όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις. Οπότε, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει με βάση την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι εμπλουτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν, δεν, δεν χτυπήθηκαν με τίποτα από τη διεύρυνση οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Άρα, επομένω, πρόκειται για μια τρομομηχανή, πρόκειται για μια κινητήρια δύναμη. Αυτό είναι η διεύρυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, χωρί τι οικονομικέ δυνατότητε, το, το δυναμικό τη ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τότε η, ο κατασκευαστικό, μάλλον η, βιομηχανία, ε, της ε, Δυτικής Ευρώπης επρόκειτο να μετεγκατασταθεί αλλού, εκτός Ευρώπης. Να, βλέπετε επομένω. πόσο βόηθησε η Ανατολική Κεντρική Ευρώπη την βιομηχανία στην Ευρώπη, τη βιομηχανική παραγωγή. Και επομένω μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για τα Δυτικά Βαλκάνια τέτοια προοπτική υπάρχει. Τα Βαλκάνια επομένω μπορεί να είναι ακόμα μια κινητήρια δύναμη που να δώσει όθηση στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στη να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να προετοιμαστούν για να γίνουν μέλη της Ένωσης. Έχουμε κάποιες κοινέ αξίες, έχουμε κάποια ε, εσωτερικά προβλήματα ε, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες αρχές, ιδίως όσον αφορά την χρηστή οικονομική διαχείριση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να γίνουν μέλη της Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, να σπαστούν αυτές τις αρχές. Να γίνουν κοινωνοί λοιπόν αυτών των αξιών τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως, για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση θα πρέπει να έχουμε και εμείς ανοιχτή θέση. Θα πρέπει τα Βαλκάνια να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να σπαστούν αυτέ τι αξίε και προσωπικά είμαι πεπισμένο ότι τα προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να επιληθούν και άρα θα πρέπει και εμεί να του δώσουμε την ε, ευκαιρία. Τώρα, να δούμε τι στόχους έχουμε, τι μπορούμε να καταφέρουμε από κοινό. Όσον αφορά την Κροατία, νομίζω ότι η Κροατία μπορεί να είναι μια χώρα υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση. Απόδειξη του πώς είναι κάτι το εφικτό, το ευρωπαϊκό όνειρο σταθερότητα, προοπτική ένταξης, όλα αυτά τα οποία βοηθούν την σταθερότητα της χώρας. Τώρα, όσον αφορά κάποια σχόλια που διατυπώνονται σε σχέση με την προσχώρηση της ε, Κροατίας και συνδέουν την υποψηφιότητα με την σύνδεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σερβίας. Αυτά τα σχόλια είναι επιβλαβή και για την Κροατία και για τη Σερβία. Δεν θα πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν ε, ε, διαφορές, ε, διαφορετική, είναι, υπάρχει διομορφία σε κάθε χώρα και άρα είναι μεγάλο λάθος να γίνονται τέτοιες σκέψεις, τέτοιες διατυπώσεις. Έτσι πρόκειται για σενάρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι παρασυρώμαθα σε πάρα πολύ επιζήμιες συγκρούσεις και αναμετρήσεις ε, απόψεων. Αυτό που κάθε φορά πρέπει να ισχύει είναι να εξετάζεται η επίδοση, οι επιδόσεις της κάθε χώρας. Αυτό πρεσβεύει η Ουγγαρία. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να προχωρήσουν και το γνωρότερο να τον κλείσουν οι διαπραγματεύσει με την Κροατία. Όσον αφορά τώρα το Μαυροβούνιο, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν το νωρίτερο δυνατόν οι διαπραγματεύσει. Βέβαια και για την Κροατία το ίδιο ισχύει και είναι σημαντικό η Σερβία να χαρακτηριστεί υποψήφια χώρα και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο. Αλλιώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παράδοξο που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα. Εμείς είμεθα πολιτικοί που αναδειχθήκαμε μέσα από ελεύθερες εκλογές. Και θα πρέπει επομένω να μην θεωρούμε ότι είναι τόσο δύσκολο το να χρησιμοποιήσουμε το όνομα που διαλέγει μόνη της μια χώρα για τον εαυτό της και να μην χρησιμοποιούμε ονόματα όπως Φιρόμ, Πουγουδουμού. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της υποψηφιότητας της χώρας αυτής. Αυτό προσβεύει και η Ουγγαρία. Το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει επομένω να εξεταστεί η υποψηφιότητα της χώρας εκείνης και δεν θέλουμε να υπάρχουν εμπόδια στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη χώρα αυτή. Περί τα τέλη των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να κάνουμε το θέμα της, ε, του ονόματος, της ονομασίας. Τώρα, όσον αφορά την Αλβανία. Είναι δυνάμει και η Αλβανία είναι υποψήφια. Ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, έχουμε τα 12 κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί η χώρα. Όμω και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει νωρί και να μην αναβάλλονται περαιτέρω, διότι μια τέτοια παρέλκυση θα έφερνε λιγότερη σταθερότητα στη χώρα. Επίσης, για την Αλβανία θα πρέπει και για αυτήν τη χώρα να μείνει ζωντανή ελπίδα η ευρωπαϊκή προοπτική. Βέβαια υπάρχει εδώ το θέμα της αναγνώρισης του κοσμοπεδίου που κάποιες ε, χώρες δεν το έχουν αναγνωρίσει. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι η χώρα η οποία ίσως είναι η πιο μεγάλη πρόκληση για μας. Η χώρα τώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Προσοχή γιατί τα προβλήματα εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να δούμε πόσο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να μην εμπλακούμε και επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η Ουγγαρία είναι κοντά στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη και παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση και θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα όσα με επιτυχία έγιναν στις γειτνιάζους με την Βοσνία Ζεγοβίνη χώρας. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια θαραλέα πολιτική. Και προς τούτο θα πρέπει να συστρατευτούν όλες οι πλευρές και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Με τόλμη επομένω να ξεπεραστούν όλες οι επιφυλάξεις και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμποδίζουν την προσέγγιση. Μπορείτε πάντοτε να υπολογίζετε στην Ουγγαρία ε, για ε, αυτό το σκοπό της ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Και τώρα ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο για να κάνετε την ομιλία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι πρώτα πρώτα, θα ήθελα να σας πω πόσο χαίρομαι που παρίσταμε σε αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση που αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια σήμερα και τον Μάιο του 2008 είχα συμμετάσχει σε μια συνάντηση ακριβώς σαν την σημερινή και σήμερα βλέπω εδώ να παρίστανται και άλλοι που είχαμε βρεθεί τότε σε εκείνη την εκδήλωση σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, ε, σε κρατημέλη, προσπαθούμε, συζητούμε αυτά τα οποία συζητούνται και στα Εθνικά Κοινοβούλια και η επιτυχία εξαρτάται από το πόσο θα συνεργαστούμε επιτυχώς μαζί σας. Συνεργασία χρειάζεται με τα Εθνικά Κοινοβούλια, χρειάζεται να συνεργαστούν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Επομένω, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα πρέπει να ανταλλάξω απόψη μαζί σα για την περαιτέρω διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ορθώς θεωρήθηκε η διεύρυνση σαν την πιο πετυχημένη πολιτική που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θα το διορθώσω και θέλω να πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Δημοκρατία, σταθερότητα, ευημερία φέρνει. Παντού στην Ευρώπη. Έτσι, ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή οικογένεια που γεννήθηκε από έναν πάρα πολύ επώδυνο τοκετό τους πολέμους του 20ου αιώνα και οπότε ακόμα και ε, προσβλέπουν προς εμάς, προς αυτή την ε, ε, υπόσχεση και ακούσαμε τι είπε ο κύριος Σόρμπαν προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο θα πρέπει να συγχαρούμε για το πόσο έχει στρατευτεί για την περαιτέρω διεύρυνση, για το πόσο και προσωπικά ενδιαφέρεται και ασχολείται με την Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως, η ενοποίηση ποτέ δεν θα έχει συμπληρωθεί, ολοκληρωθεί χωρίς να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ενδιαφέρεται ε, για τις προοπτικές της ευρύτερης εκείνης περιοχής ακριβώς ε, όπως αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα του 2003 της Συνόδου της Θεσσαλονίκης και ήμουν τότε μέλος εκείνου του συμβολίου που έλαβε αυτή την απόφαση. Είμαι περήφανος γι' αυτό και άλλωστε από το 86 είχα ασχοληθεί με το πώς θα ενταχθεί η χώρα μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε και για Φινλανδία, Αυστρία, Σουηδία επίσης όσοι προς εξωτερικών και εγώ προσυπέγραψα για να γίνουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήμουν εκεί επομένως τότε που είχαμε το τελευταίο πρόσφατο τελευταίο, όχι πιο πρόσφατο, δεν το τελευταίο κύμα ε, προσχώρησης και υποψηφιωτήτων. Μόλι την περασμένη εβδομάδα είχα πάει σε Κροατία, Βοσνία, Τζεκοβίνη, Μαυροβούνιο και στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Επίση πρόκειται να πάω σε Κωσυφοπαίδιο και Αλβανία ε, τον επόμενο μήνα. γιατί πήγα εκεί, Γιατί έχει ακριβώ ανανεώσει την δέσμευσή τη για την περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και έτσι επιβεβαιώνουμε το ότι κάθε μέρα καταβάλουμε κοινέ προσπάθειε. Το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προ τι χώρε αυτέ. Τους βλέπουμε σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας των Εθνών και όλοι μας είμαστε ε, μέλη μιας τέτοιας Ευρώπης και επομένως θεωρούμε ότι αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης όμως για να γίνει κανείς μέλος θα πρέπει να κάνει κάποια πορεία, κάποια διαδρομή, αλλάζει η περιοχή και θα πρέπει επομένω αντίστοιχα να κάνουν βήματα αποφασιστικά όλε αυτέ οι χώρε. Όλε αξίζουν να τα κάνουν όλα αυτά, να ε, έχουν αυτή την πετυχημένη πολιτική της ένταξης, οπότε πάντα έτσι θετικά βλέπουμε τα πράγματα και να ξεκινούμε από την Κροατία και που θα είναι θετικός καταλήτης για όλη την περιφέρεια, όλη την περιοχή η οποία θα πρέπει σταθερά να κατευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και πήγαμε εκεί και για να δώσουμε μήνυμα αλληλεγγύης, αλληλεγγύης και για ενθάρρυνση. Πάντως η κατάσταση εκεί είναι περίπλοκη. Έχουμε μπροστά μας ε, ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Μπαίνουμε στην τελική φάση για την Κροατία και αν όλα πάνε καλά μέχρι τον Οκτώβριο θα ισχύσει το ίδιο για Μαυροβούνιο αλλά και την Σερβία. Να δούμε πάντως ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ε, προκλήσεις ε, από μέχρι, ε, μέχρι Βελιγράδι θα πρέπει να δούμε πώς θα απεμπλακεί κατάσταση για Αλβανία για Βοσνία, Τσεκοβίνη, αλλά και να λυθεί το θέμα της ονομασίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει κράτος δικαίου σε όλη την περιοχή και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο ε, σας απασχόλησε στην ομάδα εργασίας όσον αφορά συνεργασία για ελευθερία, δικαιοσύνη για ασφάλεια και επίσης ευχαριστώ την Doris Σπακ και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας, ε, μας είπε για τη δουλειά των ε, ομάδων εργασίας, ε, δημοκρατικά θεσμικά όργανα, μια δικαιοσύνη που λειτουργεί, σεβασμός των δικαιωμάτων, των μειονοτήτων, όλα αυτά είναι βασικά τα οποία θα πρέπει να ε, να γίνουν και όχι μόνο να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, χρειάζονται επενδύσεις, να τονωθεί η ανάπτυξη, όμως θα πρέπει οι ξένοι επενδυτές να ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιες εγγύσεις από δικαιοσύνη, ε, από δημόσια διοίκηση έτσι θα πρέπει αποφασιστικά να προχωρήσουν προς κάποιες μεταρρυθμίσεις και έτσι να αντιμετωπίσουν τις σχετικές προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή προοπτική θα βοηθήσει στη σταθερότητα, εκδημοκρατισμό, ε, σε ανάπτυξη αυτών των ε, χωρών, των υποψηφίων και των ενδυνάμει υποψηφίων. επομένω. έτσι ε, θα υπάρξει ευημερία για όλους τους πολίτες και έτσι θα έχουμε μια βιώσιμη πορεία ένταξης και αξιόπιστη. Όπως και και στο Σαμπόρ της Κροατίας θα πρέπει να ε, βασιζόμαστε σε αξιοπιστία, σε αμοιβή εμπιστοσύνη. Όλο ο κόσμο να ξέρει ότι μόλι μια χώρα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πάνε να πει ότι μπαίνουν σαν μέλη, ισότιμα, πλήρη. Άρα, δεν είναι η ένταξη μια γραφειοκρατική διαδικασία συμπλήρωση ενό εντύπου. Πρόκειται για έναν μετασχηματισμό. Πρόκειται για μετασχηματισμό όλη τη χώρα. Πρόκειται για ευκαιρία εξυγχρονισμού όχι μόνο του κράτους αλλά και όλες τις κοινωνίες της χώρας. Και όλα αυτά βγαίνουν μόνο μέσα από μια συνένεση όλου του πολιτικού φάσματος για τις αλλαγές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα. Άρα και οι χώρες των Βαλκανίων να ξέρουν ότι πάντοτε θα είμαστε δίπλα τους, μπορούν να υπολογίζουν σε πολιτική, οικονομική, ε, αλληλεγγύη και υποστήριξη. Όχι μόνο λόγια. Ήδη υπάρχει τέτοια υποστήριξη και ήδη έχουμε κάνει τη διαφορά σε πολλές υποψήφιες χώρες. Συγκεκριμένη έκφραση τούτου είναι η οικονομική ενίσχυση, η προενταξιακή. Μέχρι το 2013 έχουμε δώσει 11,5 δις ευρώ για θεσμικά όργανα, ανθρώπινους πόρους, ε, ανάπτυξη στην περιφερειακή αλλά και της υπαίθρου και για την διασυνοριακή συνεργασία. Και έτσι, για να είμαστε πιο κοντά, καταργήσαμε την βίζα των διαβατηρίων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδίω για τους νέους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις κοινωνίες των χωρών αυτών. Παρ' όλα αυτά, παρά την αρρωγή προς αυτές τις χώρες, χρειάζεται να σημειωθεί πρόοδος και να γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται ηγεσία δυναμική, αμοιβαίο συμβασμό και θέληση συνεργασία. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που κάνουν τα Δυτικά Βαλκάνια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γυρίσει η σελίδα σε σχέση με το δύσκολο πρόσφατο παρελθόν. Πάμε για μια κουλτούρα συμβιβασμού, συνένεσης, αξιοπρέπειας. Δεν είναι αδυναμία η συνένεση. Αντίθετα, οποίο μπορεί να συμβαστεί, γίνεται ισχυρότερος. Ε, έγινε και αυτή η ομάδα εργασία σα για του πολίτε, για την, ε, ε, για την πολυμορφία, την πολιτιστική. Κοίταξτε, ποτέ καμία χώρα δεν έχασε την ταυτότητά της την μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο γίνεται. Όταν ερχόμαστε πιο κοντά, τότε αναδεικνύεται ο σεβασμός, η πολιτική μας ταυτότητα. Όχι, δεν ε, έχουμε... Αυτό δεν είναι μια δυναμία, απλώς χρειάζεται με κοινή θέληση να προχωρούμε. Και όπως είπα και με του ομιλητέ την περασμένη εβδομάδα, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται από το αντίστοιχη πολιτική βούληση, θα πρέπει όλα τα κόμματα με, με ενότητα να συγκλίνουν προς τα εκεί. Αυτό χρειάζεται εθνική συνένεση για να υπάρξει πρόοδο προ την ε, ένταξη. Αμοιβαίο σεβασμό και συμβιβασμό. Επομένως, Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω και σε εσά και όχι μόνο στι κυβερνήσει. Ούτω ώστε να προχωρήσουμε προ αυτή τη συνέντευξη που τη χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα επιδείξετε την θέληση που χρειάζεται για να πετύχετε. Και από αυτά που είδα στο ταξίδι μου στα Βαλκάνια επιβιώθηκε αυτό το οποίο πιστεύω. Όλοι συμφώνησαν ότι έτσι θα προχωρήσουμε προς περισσότερη ευημερία. Και μου είπανε το μόνο στο οποίο συμφωνούμε όλοι, όλα τα κόμματα είναι η ένταξη, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όμως, καλό αυτό, αλλά δεν αρκεί, χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις πάνω σε βάσει συνένεση και η αλήθεια είναι ότι σε πολλέ αυτέ τι χώρε έχουν προχωρήσει περισσότερο από άλλε. Επομένω, χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται να υπάρχουν ε, κάποιοι στόχοι στρατηγικοί που να τηρηθούν, αλλά πρόκειται όμω για έναν ε, στόχο ε, που έχει στρατηγική σημασία, ιστορική σημασία. Θα μην χαθεί αυτό το τρένο και εγώ το επανέλαβα ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα, ένα στόχο ιστορική σημασία. Ο Ζωζάν Μονέ, ένα από του πατρέ τη Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είπε ότι όλοι έχουμε φιλοδοξίες και θα πρέπει να έχουμε φιλοδοξίες και να γίνουμε κάτι και για να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνονται μεταρρυθμίσεις. Οπότε οι χώρες αυτές θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό μια φιλοδοξία, θα πρέπει αυτή η φιλοδοξία να ε, πραγματοποιείται, να, να, να, να λαμβάνει σάρκα και οστά με πράξεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να συμπαρίσταται αυτέ τι χώρες. Μπορείτε να υπολογίζετε στην αλληλεγγύη μας, στην ενθάρρυνσή μας, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον σας είναι κοντά μα σαν μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Μπαρόσο για αυτή την ομιλία σας και τώρα ήρθε η ώρα για τη συζήτηση κυρίες και κύριοι με τη συμμετοχή της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κανόνες της συζήτησης θα είναι οι εξής. Αυτοί που ακολουθήσαμε και χτες θα είναι. Δηλαδή, αν επιθυμείτε να μιλήσετε, Παρακαλώ να συμπληρώσετε το έντυπο που σας έδωσαν, που έχει κάθε αντιπροσωπεία, για να ζητήσετε να παρέμβετε. Θα ετοιμάσουμε μετά εμείς έναν κατάλογο παρεμβάσεων, ομιλητών, βασισμένοι σε αυτά τα έντυπα που θα μας δώσετε συμπληρωμένα. Και ο χρόνος για κάθε παρέμβαση θα είναι τρία λεπτά θα μπορείτε να βλέπετε το χρόνο που περνάει εκεί στην, στην οθόνη και παρακαλώ να σέβεστε αυτό το χρονικό όριο. Σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εφαρμόσουμε και τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από μια παρέμβαση τριών λεπτών θα υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ευρωβουλευτής να υποβάλει ερώτηση, έχει στη διάθεσή του 30 δευτερόλεπτα και η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πάλι. Και τώρα ήρθε η ώρα να συμμετάσχετε εσείς, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ο κύριος Μπουστινάρου, που θα είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Είναι εκτός μικροφώνου ο κύριος Μπουστινάρου, δεν τον ακούμε οι διερμηνείς. Δυστυχώς πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο, δεν ακούμε τίποτα κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Ορμπάν. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε κάτι διαδικαστικό. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, εδώ και αρκετούς μήνες σας έστειλα μια επιστολή. Εκεί σας ενημέρωνα για τη δήλωση που έγινε κατά του προσώπου μου, που είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από την κυρία Ζωζεφίνα Τοπάλη που είναι πρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου που είναι εδώ σήμερα. Η κυρία Τοπάλη με κατηγόρησε στις 24 Φεβρουαρίου στο Ελβανικό Κοινοβούλιο από τη θέση της Προέδρου του Κοινοβουλίου ότι είμαι ρατσιστής, αντιαλβανός και διεφθαρμένος. Επίσης προσέθεσε ότι πολέμησα κατά του καθεστώτος απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίων στην Αλβανία. Η δήλωση αυτή της σχεση το πάλι είναι αβάσιμη και είναι σοβαρή και απαράδεκτη. Προσβάλλει όχι εμένα και την αξιοπρέπειά μου, αλλά καθώς και τα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε το θέμα αυτό περίπου εδώ και ένα μήνα. Γνωρίζω ότι και εσείς κύριε Πρόεδρε, από την ψηλή θέση που κατέχετε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσπαθήσατε επανειλημμένα με διπλωματικό διπλωματικές, διά, διπλωματικές διάβλους αλλά όχι μόνο αυτές να πείσετε την κυρία Τοπάλη να αποσύρει τις κατηγορίες της. Δεν θέλω να ξεκινήσω εδώ μια συζήτηση, είναι κάτι άσκοπο εξάλλου διότι εστιαζόμεθα επί σημαντικότητα του θέματος που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ήπειρό μας στο σύνολό της. Ήθελα όμως να το αναφέρω αυτό στην πολύ σημαντική αυτή ε, συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ. And σας ευχαριστώ πολύ. Έχω, βλέπ, βλέπουμε δύο γαλάζιες κάρτες στην αίθουσα. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε όσον αφορά αυτό που υπόθηκε μόλις τώρα. Υπέγραψα, υπέγραψα σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία για ένα σύντομο σχόλιο. Μετά θα είχα μια ερώτηση προς τον κύριο Όρμπαν, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τοπάλη σήκωσε γαλάζια κάρτα. Έχετε λοιπόν την, ε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μποστινάρου ότι αυτά που, είπαν είναι εντελώς, αυτά που είπαν είναι εντελώς άχρηστα. Δεν υπάρχει επεισόδιο το πάλι Μποστινάρου. Υπάρχει ένα Μποστινάρη που πρότεινε να, να μην επιτρέπει στους Αλβανούς να κινούνται ελεύθερα, να τους επιβάλλει ξανά ε, ε, τον περιορισμό. Και υπάρχουν 3,2 εκατομμύρια ε, και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ Ζεζεφίνα το πάλι που θεωρούν αυτή την αξιοκατάκριτη ε, πρόταση σαν αντιαλβανική ρατσιστική. Είναι ένα ρατσιστικός νόμος και κινητοποιείται από χαμηλά συμφέροντα. Υπογραμμίζω ότι τέτοιες προτάσεις, με τέτοια πρόταση, τέτοιες προτάσεις σε στυλ Τσαουσέσκου ε, χρηματοδοτούνται από κύκλους αντιαλβανικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν οποιοδήποτε προσβάλλεται από την πραγματικότητα, το σφάλμα δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε των 3,2 εκατομμυρίων Αλβανών, ούτε και της Ζωζεφίνα. Το πάλι είναι το λάθος. Θα ήθελα να ρωτήσω, ε, να ζητήσω από τους συναδέλφους να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση ή δυνατόν, σας παρακαλώ, σε αυτό το συγκεκριμένο βήμα που βρισκόμαστε και ας έρθουμε στο θέμα μας και ας συζητήσουμε ποια, πιο ουσιαστικά θέματα. Αντριουκάητες, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που παρενέβησαν, τον κύριο Όρμπαν, τον κύριο Μπαρόζο. Αυτό που θα ήθελα είναι θα ήθελα να συνοψίσω αυτές τις συζητήσεις αυτών των δύο ημερών. Είμαι πρόσωπος του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο, όλα τα κόμματα στη Λιθουανία υιοθέτησαν μια δήλωση συγχαίροντας την Κροατία για τα επιτέγματα της και ευχόμενοι όλοι να ολοκληρωθούν ε, το φθινόπωρο οι διαπραγματεύσεις, να ακολουθήσει η επικύρωση της ε, συνθήκης και ένα επιτυχές δημοψήφισμα για την ένταξή του στην Ευρώπη. Επίσης θέλουμε η Σερβία να μπορέσει να αποκτήσει το καθεστώς ε, της υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας και να ολοκληρώσει τον διάλογο η Σερβία με το Κωσυφοπαίδειο τις διαβουλεύσεις σχετικά. Επεκτείνουμε αυτά τα συγχαρητήρια προς τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, ε, και πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα βοηθήσουν τον διάλογο μεταξύ Μακεδονίας, λέει ο μιλητής, και της Ελλάδας για να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι περισσότερο ενεργά θα μπορούσε να εμπλακεί και στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη όπου θα έπρεπε να καταβάλει προσπάθειες. Η κατάσταση εγχώρια στην Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η πιο περίπλοκη πιστεύω. Και κατανοούμε φυσικά από την άλλη πλευρά ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες από πλευράς τους. Πολλές φορές ε, κατανοούμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης και τη σπουδαιότητά τους. Όλα αυτά είναι δεκτά. Θέλουμε να τονίσουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταδείξει αλληλεγγύη προς τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Και ως προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς η ανατολική γειτονία, η σχέση ανατολικής γειτονίας και η πολιτική γειτονία θα, θα έπρεπε να είναι ένα καλό παράδειγμα. Η Λιθουανία περιτριγυρίζεται από, έχει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη Λευκορωσία, Μπελαρούς, έχουμε την περιοχή του, Καλίνιν, του Καλίνιγκραντ, θύλακα της Ρωσίας. Πιστεύουμε στην ε, επιτυχία των Δυτικών Βαλκανίων. Πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να αντανακλάται η επιτυχία αυτή και για την ανατολική γειτονική σχέση και πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανατολικούς εταίρους μας. Και γι' αυτό η Λιθουανία θέλει να εμπλακεί πιο ενεργά σε αυτές τις διεργασίες. Εχθές είχαμε μια συζήτηση για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ασφάλεια και το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης ασφάλειας. Συνειδητοποιούμε απόλυτα την ανάγκη να ενταθεί η αστυνομική συνεργασία, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με Frontex. Ευελπιστούμε και έχουμε εμπιστοσύνη στη Frontex η οποία καταβάλει αποτελεσματικές προσπάθειες και πιστεύω ότι αυτό το φόρουμ, αυτό το βήμα σήμερα θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως σημαντική προώθηση ώστε να προωθούν αυτά τα θέματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για να ενδυναμωθεί η ολοκλήρωση. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Όρμπαν. Θα ήθελα λοιπόν να διατυπώσω το εξή ερώτημα. Ερωτώ κύριε, ποια είναι η άποψή σα κατά τη διάρκεια τη προεδρία σα. Δεν θα έπρεπε να ενεργοποιηθείτε περισσότερο, να καταβάλλετε περισσότερε προσπάθειε ώστε να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδο για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Κοιτάξτε συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά τους κανόνες του παιχνιδιού, τη συζητήσεως με άλλα λόγια. Εάν σηκώσετε γαλάζια κάρτα, έχετε 30 δευτερόλεπτα να υποβάλλετε ερώτηση. Εκτός της κανονικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει όταν σηκώνετε τη γαλάζια κάρτα σας. 30 δευτερόλεπτα. Και εκείνος που υποβάλλει την ερώτηση 30 δευτερόλεπτα και εκείνος που απαντά 30 δευτερόλεπτα. Και έχουμε και τις κανονικές παρεμβάσεις των τριών λεπτών. Αυτές εντάσσονται σε μια άλλη διαδικασία κυρία Αντρεκαίτης ε, αυτό έκανε θα έπαιρνε το λόγο αργότερα ήταν στον κατάλογο των ομιλητών και μίλησε τώρα αλλά δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει τώρα ο Πρωθυπουργός αν θέλετε να απαντήσετε έχετε το λόγο Σας ευχαριστώ με τη σωστή σειρά η σωστή σειρά θα έλεγα είναι η εξή. Πρώτα πρέπει να έχουμε ένα όραμα και μετά στη συνέχεια πρέπει να καταλήξουμε στην δημιουργία μια επιτυχού ιστορία και μετά να αντιμετωπίσουμε το θέμα Βοσνία Ζεγοβίνη. Ήταν σωστό αυτό που έκανε η Ουγγρική Προεδρία, πιστεύω, να ενδυναμώσει την συνεργασία για την ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων για να υπάρξει ένα όραμα για την πολιτική μα. Μετά θέσαμε ιδιαίτερη σημασία η Κροατία να μπορέσει να στεφθεί με επιτυχία επιτυχία στο εγχείρημά τη στην πρωτοβουλία τη Να χρησιμοποιηθεί ω μέσο ώστε να βρεθεί ευθυγραμμισμένη η Βοσνία Ερζεγοβίνη προς την πορεία ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ο Λόρδο Μπάουνας έχει το λόγο εκ μέρου τη ε, Βουλή των Λόρδων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που δίνετε δυνατότητα να συμβάλλω κι εγώ στην ε, συζήτηση και μας τιμά η παρουσία του Πρωθυπουργού Ορμπάν και του Πρόεδρου Μπαρόσο. Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα εδώ κατά τη διάρκεια του διμέρου κατέδειξαν ότι ανάμεσα αντιπροσωπείες είτε αυτές ήταν από τα παρόντα κράτη-μέλη είτε από τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή υπεποίθηση ότι το μέλλον των Βαλκανίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε θαρρυντικά λόγια για τα εφιστάμενα προγράμματα, την υποστήριξη και τη συνεργασία που υπάρχουν και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Όμω, θα πρέπει να τονίσω ότι οι μεταρρυθμίσει που είναι δύσκολε για τον κόσμο, δύσκολο να εφαρμοστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε απογοητεύσει, εάν δεν ιδωθούν ω πρόοδο προ τον τελικό στόχο. Οπότε δεν υπάρχει υποκατάστατο, όπω είπα και χθε, κύριε Πρόεδρε, α για ουσιαστική πολιτική δραστηριότητα και αποφασιστική προσπάθεια που θα εξασφαλίζει το ότι η πολιτική βούληση και η επιθυμία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να δει την διεύρυνση στα Βαλκάνια είναι υψηλά στην ημερήσια διάταξη κάθε Προεδρία. Βεβαίω, παραδέχομαι τη δουλειά που έκανε η Ουγγρική Προεδρία, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να εξακολουθεί να γίνεται αυτή η προσπάθεια και σε επόμενε Προεδρίε. Θα πρέπει να συμβιβαστούμε σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούμε να ισχύουν για να γίνει μια χώρα μέλο, αλλά θα πρέπει δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετη η προθεσμία θα τίθεται, αλλά θα πρέπει να πληρούνται κάποιε προδιαγραφέ. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Γεγονότα αλλού δεν θα πρέπει να μα κάνουν να παρεκκλίνουμε την προσοχή μα σε αυτόν τον τομέα και για αυτή την περιοχή που είναι αναπόσπαστο τμήμα τη Ευρώπη και κάτι εκρεμέ, μια εκκρεμότητα. Θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα παντού ταυτόχρονα. Και εγώ προσωπικά καλωσορίζω την στεναρή ρεαλιστική άποψη που εξέφρασε ο Πρωθυπουργό Ορμπάν σήμερα το πρωί. Η προτεραιότητά μα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στοχευμένη βοήθεια για την καταπολέμηση τη διαφθορά εγκληματικότητα και ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα και την επιβολή του κράτου δικαίου. Και εντό αυτή τη προτεραιότητα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Κροατία θα μπορέσει να κλείσει το κεφάλαιο για το δικαστικό κλάδο και να επιταχυνθεί και να προχωρήσει μάλλον στην ενταξιακή διαδικασία. Και θα πρέπει να γίνει πολιτική προσπάθεια μεγάλη για να, για να γίνουν συνταγματικέ αλλαγέ στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η χώρα αυτή δεν θα ολιστήσει ξανά στην αστάθεια. Ε, και τέλο, σοβαρή προσπάθεια να βοηθηθεί ε, να επιλύθει το πρόβλημα τη ονομασία του ΦΥΡΟΜ μεταξύ Ελλάδα και ε, Μακεδονία, λέει είναι πολύ σημαντικό για να ανοίξει ο δρόμος για την υποψηφιότητα τη χώρα. Αυτά είναι θέματα που τακτικά θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων του Συμβουλίου για να δοθεί όθηση στη δουλειά που ήδη γίνεται και στο πνεύμα συνεργασίας στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα Ράνο Κρυβοκάπιτς εκ μέρους του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρος ότι ο εξοπλισμός είναι στα επίπεδα του, στο, ανταποκρίνεται στο ύψος του Μαυροβουνίου και θα μπορούσατε να με ακούσετε. Ευχαριστώ. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι στο επίκεντρο τα Δυτικά Βαλκάνια των προσπαθειών των επικεφαλής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ κύριε Μπαρόσο που ε, με, ήρθα να επισκεφθεί, θα μιλήσω τέσσερις μητρικές μου στις γλώσσες κροατικά, μαυροβουνικά, σλοβενικά, βοσνιακά, ταυτόχρονα. Αστό. Αξιότιμη. Τι είναι αυτό Είναι μεγάλη επιτυχία και θέλαμε πάντα να αποσαφινιστούν αυτά τα ερωτήματα, ερωτήματα τα οποία οδηγούν σε μεγάλες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήματα που δείχνουν και τις αδυναμίες, τις αδυναμίες της περιοχής μας νόμος και δίκαιο και ένωμη τάξη και ηθαγένεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε τις δικές της βάσεις για τα δικαστικά θέματα ως θεμέλια. Μας προσέφερε αυτά τα θεμέλια ώστε να μπορέσει να επιβληθεί η δικαιοσύνη. Για να επιβληθεί η δικαιοσύνη πρέπει να ε, ε, επικρατήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο δημοκρατίας, δημοκρατικού καθεστώτος πρώτα. Και δεν υπάρχει διερμηνία, ερωτά ο μιλητής. Mm. Ναι, ίσως οι τέσσερις αυτές γλώσσες δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητές, γι' αυτό συνεχίζει ο μιλητής, λέει, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Υπάρχει διαρμηνία. Uh, Και πάλι η εγκληματικότητα τώρα συνεχίζει ο μιλητής η εγκληματικότητα μετά τον πόλεμο αποδυνάμωσε ιδιαίτερα τις χώρες μας το οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Από κοινού να διασφαλίσουμε ότι τα Βαλκάνια θα είναι μια περιοχή όπου σταθερότητα και το δίκαιο θα επιβληθεί. Η δημοκρατία είναι η συνεισφορά για να επιτευχθούν αυτά. Ε, η επιβολή αυτών των αρχών ξεκίνησε με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δίκαιο και νόμος πρέπει να επιβληθεί. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και χάρη σε αυτήν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι διαπραγματεύσει για την ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτό το πρίσμα πρέπει και μπορούν να συνεχιστούν. Η ανάπτυξη και η οικοδόμηση τη κοινωνία των πολιτών στη συνέχεια. Για να καταφέρει μια χώρα να είναι ε, με σωστό τρόπο να κυβερνάτε πρέπει να μπορέσουν όλα τα τμήματα να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για μας. Παράγοντας συνοχής. Αφορά την ζωή μας, την ιδιωτική μας οικονομική κοινωνική ζωή. Και γι' αυτό η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυνατότητες για την ολοκλήρωση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικές υποθέσεις. Είναι όμως αναγκαίο να επικρατήσουν οι όροι και προϋποθέσεις εκείνη και εκείνες που τα εθνοτικά και θρησκευτικά τμήματα θα τα δίνουν ως τμήματα μόνο ενός συνόλου. Δεν μπορούν αυτά η θρησκεία δηλαδή και αυτές οι παραδόσεις να είναι εθνοτικές παραδόσεις να είναι το μόνο θεμέλιο του έθνους μας. Η πτυχή της ολοκλήρωσης και του ενιαίου συνόλου είναι αναγκαία συνιστόσα και όλα αυτά τι καταδεικνύουν. Καταδεικνύουν ότι όταν και αν στα Δυτικά Βαλκάνια θα μπορέσει να επικρατήσει η εθνοτική αρμονία, η, η συμβίωση ειρηνική και η κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων θα έχουμε προχωρήσει συνένεση και συνεννόηση και όχι συγκρούσεις. Το Μαυροβούνιο είναι ακριβώς μια τέτοια χώρα. Κατάφερε να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας να το ε, διεκδικήσει και να το κατακτήσει. Είναι δική μας ε, επιθυμία η Κροατία να μπορέσει το δυνατόν, είναι η επιθυμία μας η Κροατία να ενταχθεί το δυνατόν γοργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποτελέσει υπόδειγμα, πρότυπο για μας και να είναι πλήρη ε, υπό την πλήρη ιδιότητά της ε, η χώρα μας το Μαυροβούνιο να μπορέσει ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Θέλουμε να ανήκουμε και, και εμείς αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο μιλητής είναι ο Ρίχαρτ Χόρτσικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Μπαρόσο, Πρωθυπουργέ Ορμπάν, Πρόεδρος τη Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία τη σημερινή διάταξη Δυτικά Βαλκάνια και κάποια σχόλια έχω για την Ουγγρική Προεδρία. Κύριε Πρόεδρε, τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να είναι το τμήμα τη Ευρώπη και το μέλλον τη Ευρώπη. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρί το άλλο. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όχι πρόβλημα, αλλά δυνατότητα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό μου στην αξιοσημείωτη ομιλία του. Και πρέπει να εφαρμόζονται κοινέ αξίες, είναι δυνατότητα αυτή και να δοθεί ευρωπαϊκή προπτική για κάθε μέλος, κάθε χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι προς όφελος όλων μας θα πρέπει να αποσταλεί σαφές μήνυμα σήμερα. Σκληρή δουλειά αφοσίωση στις ευρωπαϊκές αξίες όπως το κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα όπως η απελευθέρωση από τις θεωρήσεις διαβατηρίων, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, ισχυρή Ευρώπη είναι το σύνθημα της Προεδρίας μας. Η ισχυρή Ευρώπη αφορά τα τολμηρά βήματα. Πρέπει να γίνονται όταν απαιτείται. να χρειάζεται ισχυρή οικονομία η οικονομική διακυβέρνηση σχετίζεται με αυτά τα θέματα για να εξασφαλιστούν τα προαπαιτούμενα, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταποκριθεί στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που θα πρέπει να ξεπεραστεί. Το να γίνει η Ευρώπη ισχυρότερη από ό,τι πριν από ένα εξάμεινο. Αυτό είναι ο βασικό μα στόχο. Γι' αυτό εστιάζεται η Ουγγρική Προεδρία επί στοιχείων της απάντησης που θα βρει η Ευρώπη για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Κάτι που ήταν εντός των ευθύνων της εναλλασσόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου. Υπάρχει συνεργασία με τον κύριο Βαν Ρομποέ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σε εφαρμογή του μακροοικονομικού συντονισμού και του σχετικού κύκλου, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ένα πακέτο έξι νομοθετικών προτάσεων που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης είναι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος Ουγγρική Προεδρίας. Ήδη έχουμε κάποια επιτυχία, αλλά θα πρέπει να εξακολουθήσει η προσπάθεια για να πετύχουν τους στόχους. Κύριε Πρόεδρε, η Ουγγρική Προεδρία εργάζεται σκληρά. Είναι βασικός και αξιόπιστος εταίρο και με τα να κινηθούμε όλοι μαζί για να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον που θα συμπλαμβάνει τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Ταμπάτζη, εκ μέλους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ Όρμπαν, Πρόεδροι, κύριοι Μπούσεκ και Μπαρόζο, θα έλεγα ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την Ουγγρική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε σεβασμό για τη διοργάνωση αυτής της ε, ε, συνεδρίασης. Σε πολύ σωστή χρονική στιγμή και συγκυρία γίνεται αυτή η συνάντηση. Διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια επιβράδυνση όσον αφορά την ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Μετά τις ε, μαζικές διευρύνσεις ε, το 2007 υπάρχει μια κόπωση όσον αφορά τη διεύρυνση από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχουν μηνύματα για μια άλλη κόποση στην οποία θα αναφερόμουν ως κόποση της ένταξη ή προσχώρησης. Είναι κάτι επικίνδυνο αυτό όμως. Ελοχεύουν κίνδυνοι εδώ. Το να είναι κανείς ε, ε, μέλος, η ιδιότητα κράτους ε, μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προοπτική περνάει πια στο απότερο μέλλον για πολλά κράτη. Σε σχέση με τα ωφέλη τα οποία θα μπορούσαν να αποκομίσουν η προοπτική αυτή φθήνει. Και υπάρχουν έτσι και προσχήματα για κάποιους όπως στη Μακεδονία λέει ο μιλτής, να αναβληθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ή να υπάρξει η προσπάθεια σε σχέση με τη συμφιλίωση με γειτονικές χώρες να αναβληθούν ή να κολυσιεργούν, ε, να κολυσιεργούν όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων. Σε σχέση με την ε, ε, πολιτική οικογένεια, δεν είμαι μέλος αυτής της πολιτικής οικογένειας όπως ο κύριος Όρμπαν, όμως μπορώ να εκτιμήσω τα όσα έχουν γίνει από την Ουγγρική Προεδρία για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την Κροατία σε ανώτατο επίπεδο, ώστε να αποκτήσει σάρκα και ωστά η προοπτική ένταξη αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επίσης και οι διαπραγματεύσεις με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει διστακτική ε, αντιμετώπιση σε σχέση για παράδειγμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μπορούμε να ε, καλύψουμε αυτές τις, αυτή την απόσταση στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ρωτήσω να ε, ζητήσω από την ανακυκλούμενη Προεδρία να αναλώσει τους επόμενους μήνες που έχει στη διάθεσή της ακόμα ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάσει τι θα μπορούσε να γίνει να ευδοκιμήσουν οι στόχοι που εκκρεμούν ακόμα θα πρέπει αυτός ο, ο θύλακας να μπορέσει να γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν προετοιμάσουμε ένα πακέτο σφαιρικό και συνολικό στο οποίο θα εμπλέκεται στο πακέτο αυτό και στις πρωτοβουλίες το ιδιωτικό κεφάλαιο, αν δεν κάνουμε μια τέτοια κοινή προσπάθεια σε ένα πακέτο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αυτή η κόπωση ένταξης ή προσχώρησης θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Θα διευρυνθεί η κόπωση αυτή, ο χωρεσμός και θα πρέπει να μπορέσουμε να επιλύσουμε προβλήματα γυτνίασης και προβλήματα εθνοτικά. Δεν είναι δυνατόν να αναμείνουμε μετά την προσχώρηση των χωρών αυτών για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Να θυμηθούμε τι έγινε σε σχέση με τη Σλοβακία αφού είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υιοθέτησε το νομοθέτημα σε σχέση με την γλώσσα έναντι των Ούγγρων και αρκετές ε, χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμα τα δικαιώματά τους. Διακόπτεται ο μιλητής από τον Πρόεδρο. Ευχαριστούμε κύριε. Η ε, κυρία Ζωσεφίνα Τόπαλη θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ πολύ αυτή τη μειχτή κοινοβουλευτική ε, σύνοδο και τη συνομιλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τα Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων. Και στόχο είναι πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη με τη συμμετοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλε τι κοινοβουλευτικέ ομάδε και την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών που υπερψήφισαν το καθεστώ απελευθερώσεω των θεωρήσεων διαβατηρίων για του Αλβανού πολίτε πέρσι. Ήταν μια τίμια εκτίμηση της τεραστίας πρόοδου που έχει πετύχει η Αλβανία κατά τα τελευταία χρόνια Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έκανε προσπάθειες για να υποστηρίξει την Αλβανία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ε, στην προσπάθεια ε, της ένταξης. Και σαν πρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για την αλληλεγγύη που έδειξε απέναντι στα Βαλκάνια εν γέννη και έναντι της Αλβανίας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Όπως γνωρίζετε η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και για να είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Αλβανία έκανε μεγάλη πρόοδο, τεράστιες μεταρρυθμίσεις, δραματικές μεταμορφώσεις Αν δείτε ε, εδώ και 20 χρόνια που ήταν η Αλβανία και που είναι σήμερα, βλέπετε ότι έκανε, κατάφερε να κάνει τα περισσότερα η Αλβανία σε συντομότερο χρονικό διάστημα όσον αφορά την οικονομία. Τώρα που έχουμε ένα τσουνάμι οικονομικό χρηματοπιστωτικό σε όλο τον κόσμο, η Αλβανία πέρσι είχε 4% οικονομική ανάπτυξη. Το τελευταίο τετράμινο πέρσι Είχαμε 5% οικονομική ανάπτυξη. Είχαμε ένα χρέος 59%. Το μειώσαμε κατά άλλα 2% κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Έχουμε 3,5% έλλειμμα, πληθωρισμό υποέλεγχο, 62% αύξηση των εξαγωγών. Οπότε νομίζουμε ότι στην πραγματικότητα η Αλβανία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχαμε τεχνητά προβλήματα που δημιούργησαν κάποιοι. Αυτές είναι οι προκλήσεις μιας δημοκρατίας. Ξέρουμε, δεν ήταν ευτυχής ιστορία της χώρας μας. Πάντα σαν Αλβανοί ήμασταν κάτω από την εγκληματικότητα ή υπό ε, εισβολές υπό πόλεμο. Και τώρα όμως αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη και χρειαζόμαστε οι άλλοι να είναι τίμοι απέναντι στους Αλβανούς. Οι Αλβανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα μήνυμα να στείλουμε. Έχουμε Σιήτες, Σουνίτες, Ορθόδοξους και Καθολικούς στην Αλβανία. Τέσσερις θρησκείες και ζουν αρμονικά και θα πρέπει να το δουν οι άλλοι σαν μοντέλο. Αυτό και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Δεν θέλω να είμαι αγενής με κανένα τρόπο, αλλά θα πρέπει οι αγορητές να τηρούν το όριο, το χρονικό το οποίο έχει δοθεί για τις παρεμβάσεις τους. Ο επόμενος είναι ο Λόρδος Τέβεσον από την Ανοβούλη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστώ. Παρακολουθώντα τι ε, παρεμβάσει σήμερα που ήταν εξαιρετικέ από τον Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, εξαιρετικέ στην πρακτική του ε, μορφή και τόνο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνόδου εθνικών ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτών που με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων σε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα προφανέ λόγω τη απουσία. εξετάζοντα. Του ε, τους καταλόγους παρουσίας των Εθνικών Κοινοβουλίων, εννέα κράτη-μέλη απουσιάζουν δυστυχώς. Από εκείνους που απουσιάζουν βλέπουμε την αντιπροσωπεία σε σχέση με τη Γερμανία τη μεγαλύτερη χώρα και μεγαλύτερο δωρητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε και σε σχέση και με τους όσους παρενέβησαν βλέπουμε λίγους εθνικούς βουλευτές να παρεμβαίνουν από την Βόρεια ή την Δυτική Ευρώπη. Μεγάλη αισχύνη αυτή ε, σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Είχαμε και Σουηδούς, όμως βλέπουμε ότι απουσίαζαν ε, οι άλλοι από την Βόρεια και, Κεντρική Ευρω... και ε, Δυτική Ευρώπη. Θα ήθελα σε σχέση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, συγχαίροντάς τον για την εξαιρετική του προσφώνηση, να ρωτήσω πώς θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε τους άλλους μεγάλους παίκτες σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, υποψιάζομαι ότι σε σχέση με την έλλειψη ενδιαφέροντος σε σχέση με εθνικά κοινοβούλια που απουσιάζουν εδώ σήμερα ίσως θα υπάρξει και κυβερνητική έλλειψη ενδιαφέροντος ε, για αυτή την προοπτική. Αυτό που είναι σαφές για μένα ως ε, εκπρόσωπο της Δυτικής Ευρώπης είναι ότι τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν εθνοτικά και άλλα ε, στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον αυτών των χωρών και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εμπλέκονται τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά έχουν έχουν βαρύνοντα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία να γίνει αυτό. Και δεν είναι μια λέσχη συζητήσεων, αλλά θέλουμε να, γίνουν, να ακολουθήσουν δράσει και με τι δράσει αυτέ να ενταχθεί αυτή η περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ντόρις Πακ παρακαλώ στη συνέχεια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα δύο πράγματα να πω πρόεδρε. Πρώτον πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει στα ε, Ηνωμένα Έθνη το θέμα της ε, ονομασίας ε, μεταξύ Μακεδονίας λέει ο Μιλίδρε και Ελλάδας να επιληθεί μόνο από τα Ηνωμένα Έθνη. Έχουν από πλευράς Μακεδονίας παρακολουθεί πολλά πράγματα σε σχέση με το πρόβλημα της ονομασίας. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί, ίσως έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Να υπενθυμίσω δεύτερο ότι στη Βοσνία Ζεγοβίνη που όπω προανέφερα από το Οκτώβριο δεν έχει πλέον ε, τα αναγκαθεσμικά όργανα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεωρήσουμε ότι ευθύνη μας είναι να προχωρήσουν τα πράγματα για τους πολίτες εκεί. Δεν ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες να υποχρεωθούν οι πολιτικοί εκεί να θυμηθούν το έργο τους ποιο είναι. Έχουν εκλεγεί για τη νέα γενεά, να δουλέψουν για τη νέα γενεά, για υποδομέ για καλύτερη εκπαίδευση και παιδεία, για θέσεις εργασίας. Κανένα Κανένας όμως ε, δεν έχει υιοθετήσει μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι όλοι αποτελματωμένοι σε εθνικιστικές τάσεις. Ε, αν δεν το καταφέρνουν πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να τα καταφέρουν. Υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα να εμπλακεί περισσότερο, να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. Και σε αυτό ανήκει ότι επιτέλους και για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και το Πέδιο θα πρέπει να έχουμε πρεσβείες εκεί, πρέσβεις. Δεν γίνεται εκεί με πολλές προσπάθειες, ε, με πολλά στελέχη να καταβάλουν με προσπάθειες και να μην έχουμε πρέσβει εκεί που εκεί πέρα, εκεί κάτω πραγματικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να είναι εταίρο στι συζητήσει με του κυβερνώντες. Λοιπόν, έτοιμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο έχει εδώ και πολύ χρονικό διάστημα αυτό το αίτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε κάτι περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Να προαχθούν αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί από πλευρά κονδυλίων, αλλά η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει. Πρέπει να συνεισφέρει για το Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία. Ο διάλογο μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβία πρέπει να προαχθεί. Να έρθουν πιο κοντά οι πολίτε αυτών των δύο χωρών. Λίγο περισσότερο να προσεγγίσουν οι μεν του δε. Οι Σέρβοι στο Κωσυφοπέδιο χρειάζονται την εντύπωση ότι μέσα σε αυτό το διάλογο και εκείνοι λαμβάνονται υπόψη ότι δηλαδή σε σχέση με το κοσυφοπέδιο αναγνωρίζεται η παρουσία τους και έτσι οι δυνατότητες για τους ε, κοσυφοπέδιους να ταξιδεύουν και αυτό είναι μια ανάγκη μια αναγκαιότητα όπως και η συμβίωση μεταξύ των δύο αυτών λαών των δύο εθνοτήτων σε αυτή τη χώρα Σέρβων και Κωσοβάρων η απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων πρέπει να βοηθήσουμε η στενοπός να αντιμετωπιστεί τα διαβατήρια να γίνονται δεκτά και από την Σερβία και από τη Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να δουλέψουμε και γι' αυτό δεν μπορεί να αναβάλλεται αυτό στις ελληνικές καλένδες και να μην γίνεται τίποτα και πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καταλίν Έτσεφ από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω μερικά λόγια, λέει η κυρία Ερτσέη, για την όλη ορμή της ε, διαδικασίας που ε, καμιά φορά γίνεται αντιληπτή σε αυτή την αίθουσα, όμως τίθεται το ερώτημα κατά πόσο έχουμε αυτή την ορμή πάρα έξω. Για να υπάρχει αυτή η ορμή, αυτή η όθηση, χρειάζεται φωσίωση στο στόχο. Χρειάζεται ενθουσιασμό στη συζήτηση. Υπήρξαν στιγμές στη χθεσινή συζήτηση και στη σημερινή συζήτηση όπου αισθανθήκαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να, βρούμε μια διέξοδο. Είτε θα σπρώξουμε τώρα, θα δώσουμε τελική όθηση, είτε όχι. Πρέπει να δώσουμε μια όθηση ούτως ώστε να βοηθήσουμε να ενταχθεί η περιοχή. Διαφορετικά θα επιβραδυνθεί η διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας τους πρασίνους και στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό, λέω, το θέμα και θα στηρίξουμε την Ουγγρική Προεδρία για να επιταχύνει τη διαδικασία και η διαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης να προχωρήσει. Αυτό θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από τις επιδόσεις και την συμμόρφωση των διαφόρων υποψηφίων χωρών. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό μας για αυτά που είπε σχετικά με το θέμα. Η συμμετέχοντες, η συμμετοχή μάλλον σε αυτή την αίθουσα, παρουσιάζει, δείχνει κάποιο σκεπτικισμό που επικρατεί. Ο ενθουσιασμός έχει αντικατασταθεί από κάποιο σκεπτικισμό τελικά στον αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ποικιλομορφία πραγματικά καθημερινή ε, όσον αφορά αυτές τις χώρες ή είναι απλώς ένα πολιτικό σύνθημα. Θέλει ποικιλομορφία η Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει μια εικόνα πολύ σταθερή και ομοιόμορφη για τον εαυτό της. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Θα πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε την εκπαίδευση των παιδιών. Από πολύ μικρή ηλικία να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Είναι σημαντικό και για την περιοχή που συζητούμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμβάθυνση, διεύρυνση πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Πικυλομορφία και συζητήσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε συγκρούσεις, αντιθέτως θα πρέπει να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε οι μεν τους δε καλύτερα. Και διακόπτει ο πρόεδρος την ομιλήτρια, συνεχίζει η ομιλήτρια, θέλουμε να ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό μας να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να προωθήσει τη διαδικασία, τις διαδικασίες αυτές και τις προσπάθειες στην ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρ σήκωσε γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου απευθύνεται προς την κυρία, αλλά έφυγε. Άρα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να πεθώ στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ορμπάν, να του πω ότι ανεφερθήκατε στην ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου που αναγνωρίζεται από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Όμω, από ό,τι γνωρίζω, μέχρι πρόσφατα δεν αναγνωρίζω όλε οι χώρε την ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου. Είτε έχασα κάποιο επεισόδιο και θα με ενημερώσετε και θα με φέρετε στον καλό δρόμο ή πρόκειτο, επρόκειτο προς γενικοποίησης. Πώ να εντάξουμε μια χώρα που δεν αναγνωρίζεται από τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι το ερώτημά μου. Μάλιστα. Τώρα ο Πρωθυπουργό θα λάβει τον λόγο. Ίσως υπήρξε κάποιο σφάλμα το οποίο παρισέφρισε η σε σχέση με την παρέμβαση το ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβατική σχέση με το κοσυφοπαίδιο επειδή υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα το κοσυφοπαίδιο για να είναι σαφές το τι είπα εγώ προηγούμενα επόμενος αγορητής λοιπόν είναι ο Ευρωβουλευτή, η Ευρωβουλευτήνα κυρία Κίντεγκα παρακαλώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο αγαπητοί πρόεδροι και ε, συμμετέχοντες. Είναι η δεύτερη μέρα που συζητούμε τα θέματα ολοκλήρωσης ε, στην, προς την Ευρώπη ως την μόνη ευκαιρία αυτών των κοινοτήτων των Δυτικών Βαλκανίων ε, να μπορέσουν ε, να, να ξεφορτωθούν το βάρος, το άχθος του παρελθόντος και να πορεθούν προς την ευημερία και την ειρήνη. Και ακούσαμε επίσης ότι η Ευρώπη χρειάζεται επίσης τα των Δυτικών Βαλκανίων, σίγουρα. Από πλευράς της Ευρώπης χρειαζόμαστε μια συνεκτική, μια την συνοχή όσον αφορά την πολιτική βούληση και το όραμα. Αυτό αναφέρθηκε, αλλά επίσης είναι αναγκαίο να είμαστε πιστοί σε ευρωπαϊκές αρχές και αξίες ε, όσον αφορά ίσως και το μεγαλύτερο εφικτό βαθμό σε πιστή σε αυτές τις αρχές και αξίες. Όσον αφορά την δικαιοσύνη και την ελευθερία, θα ήθελα εδώ να τονίσω την πτυχή των μειονοτήτων και την σχέση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης που πρέπει να τηρούνται απόλυτα και όχι μόνο με βάση αρχές και αξίες και ε, νομικούς ε, όρους ε, και νομικές διατάξεις αλλά καθημερινά πρακτικά στο καθημερινό πρακτικό επίπεδο. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει συγκεκριμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες για να ενθαρρυνθούν οι εθνοτικές μειονότητες νομικά νόμιμα να μπορέσουν να συμβιώνουν η μία δίπλα στην άλλη και να γνωρίσουν και να μάθουν η μία τον πολιτισμό, τις παραδόσεις ε, τις αξίες και τις αρχές της άλλης ε, ώστε να μπορέσουν να αποδεχθούν η μία μειονότητα την άλλη να αποδεχθεί η μία μειονότητα τον, πολιτισμό και την ταυτότητα της άλλης και αυτές οι προσπάθειες πρέπει να καλύπτουν τη γλώσσα, τη χρήση των γλωσσών και τους νέους ε, στα Δυτικά Βαλκάνια που θα πρέπει να μάθουν κάτι για την ευρωπαϊκή προοπτική για αυτούς τους ίδιους και αυτό είναι ένας στόχος που αξίζει να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Φαραγκό από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την εκδήλωση και έτσι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τόσο σημαντικά γιατί η Ρουμανία έχει εμπλακεί, ενδιαφέρεται για την ε, ένταξη χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση γιατί είναι όμορες χώρες με εμάς και επίσης ε, ε βεβαίως έχουμε εδώ και θέματα Schengen έτσι θα έχουμε σταθεροποίηση, σταθερότητα στην περιοχή και αυτό μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι σημαντικό για το σύνολο τη Ευρώπη. Επίση, θα φέρει και ευημερία η ένταξη των χωρών τη Δυτική Ευρώπη. Επομένω, όλοι έχουν συμφέρον και ενδιαφέρονται για την ένταξη. Ε, και οι χώρε των Βαλκανίων και η Δυτική Ευρώπη, αλλά και ο κάθε Ευρωπαίο χωριστά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει οριμότητα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με οριμότητα τα θέματα μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης. Το δουλεμπόριο, διακίνηση προσώπων, παράνομιο, ε, το οργανωμένο έγκλημα από πάσης απόψεις θα πρέπει να ενεργήσουμε και θα πρέπει βέβαια και οι χώρες, οι υποψήφιες να τηρήσουν τα κριτήρια της ένταξης. Ξέρουμε πόσο πολύ ταραχή είναι η ιστορία των Βαλκανίων, ξέρουμε το πώς οδηγηθήκαμε στο να έχουμε συνύπαρξη στην περιοχή τόσων διαφορετικών εθνοτήτων αλλά και μειονοτήτων. Θα πρέπει βέβαια ο καθένα να μπορέσει να διατηρήσει την ταυτότητά του και θα πρέπει να αποφύγουμε τι δυσμενεί διακρίσει και θα πρέπει όλοι να απολάβουν των ίδιων δικαιωμάτων. Και οι μειώνεται όπω και η πλειοψηφία. Ε, εμείς επομένω ε, θεωρούμε ότι όλοι ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια η οποία πρέπει να ενοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Γιάκουμ Κράσνιακ. Τώρα είναι ο επόμενος ομιλητής μας. Πρόκειται από το Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, δεν είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, εδώ και 12 χρόνια η χώρα μας αισθάνεται την επιρροή, την υποστήριξη, τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, επομένως υπάρχουν και από τις δύο πλευρές και από εμάς και από εσά η θέληση της προσέγγισης. Βέβαια, θα πρέπει να ασχοληθούμε με ζήλο, με ενεργητικότητα, να προχωρήσουμε προς ό,τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε, να προσεγγίσουμε και άλλο την Ευρώπη και εσείς να μας βοηθήσετε αντιστοίχω. Ξέρετε ότι έχουν πάρα πολλούς νέους στη χώρα, οπότε θα πρέπει να ποντάρουμε στις ε, ακάματες προσπάθειες και της νέας γενιάς. Επομένως χρειάζεται το όραμα, αλλά χρειάζονται και συγκεκριμένες προσπάθειες, συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει σε αυτή την πορεία να υλοποιηθούν. Και για όλα αυτά επίσης υποστηριζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε απομονωμένοι μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Δεν θέλουμε να καταργηθούν ε, οι θεωρήσεις διαβατηρίων εάν δεν είμαστε συνεπείς και εμείς στις προς ταχθήσεις προϋποθέσεις. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, στρατηγική που προβλέπεται και να φτάσουμε τελικά στην ε, κατάργηση αυτών των θεωρήσεων. Μιλούμε για πέντε χώρες μέλη που ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει τη χώρα μας. Αυτό δεν βοηθάει την διαδρομή μας. Να αναγνωριστεί η χώρα μας. Μια χώρα που με τους γείτονές της συμπορεύεται προς την κατεύθυνση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής σας. Ο κύριος ε, Μποστινάρου, Ευρωβουλευτής από την Ουρμανία, έχει τον λόγο τώρα. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, να σα πω για κάποια από αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί, κάποια θέματα τα οποία κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα-πρώτα, ήταν πάρα πολύ θετικά τα όσα είπε στην ε, εισήγησή του ο κύριο Όρμπαν, ε, ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, ε, και α ανήκουμε στη διαφορετική πολιτική οικογένεια, θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα είναι πολύ κοντά οι θέσει μα. Είναι πάρα πολύ α, έντονο σήμερα το ότι η, η, η Δύση έχει κουραστεί ε, έχει την κόπο της διεύνησης και η Ανατολή έχει την κόποση της ε, αναμονής. Δεν είναι αυτονόητη η ειρήνη. Ε, δεν, δεν είναι κάτι το, το, οποίο θα, θα πρέπει να το να ότι μόνο το ρυθμίζεται γιατί αν προχωρήσουμε προς την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων τότε θα έχουμε πετύχει την ειρήνευση και την ειρήνη. Επομένως χρειάζεται να υπάρχει πολιτική συνένεση σε όλο το πολιτικό φάσμα όσον αφορά την διεύρυνση προ τα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως, κάτι το οποίο μας δίδαξε η προηγούμενη διεύρυνση για Ανατολική ε, προς Ανατολική Ευρώπη είναι το, το ότι υπήρχε ευρεία συνένεση. Εάν υπάρχει αντί για τη συνένεση αντιπαράθεση για τα Βαλκάνια, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Τότε απλά θα έχουμε ε, παραβλάψει αν όχι καταστρέψει τις προοπτικές. Επομένως, αυτό που θέλω να σας συμβουλεύσω ως φίλος είναι φροντίστε να σχηματιστεί συνένεση. Γι' αυτό το ένα, το εθνικό συμφέρον, το εθνικό ζήτημα, την διαδικασία τη διεύρυνση. Επίση, για να κάνουμε να τλήσουμε συμπεράσματα και από την άλλη διεύρυνση, τη διεύρυνση προ Ρουμανία και Βουλγαρία. Χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση διοικητική. Έτσι, να μπορέσουμε να κάνουν τη διαδρομή τη ένταξης διότι αν δεν υπάρχει κάποια με τέτοια μεταρρύθμιση αποτελεσματική τότε οι χώρε σας δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν την απορρόφηση των κοινωτικών κονδυλίων ούτε και των προενταξιακών κονδυλίων. Να, τι θα πρέπει να κάνετε για αυτή την περίοδο πριν την ένταξη. Ξεκινήστε τώρα και να έχετε κατά νου ότι αυτός ο σημαντικός στόχος είναι που μπορεί να σας απασχολεί τώρα για να δούμε τι μεταρρυθμίσεις να γίνουν και όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα στα Βαλκάνια. Είναι φανερό ότι θα πρέπει το, σχετικό ε, διάστημα να γίνει. Θα πρέπει να αποσυνδεθούν τα πολιτικά κόμματα από τη διαπλοκή με τις επιχειρήσεις και από την άλλη μεριά ε, να ξεκαθαριστεί το πώς γίνεται η χρηματοδότηση των κομμάτων, διότι η, διαπλοκή και η διαφθορά δεν αφορά μόνο τα Δυτικά Βαλκάνια. Γίνεται παντού. Γίνεται παντού όπου το χρήμα βρίσκεται κοντά ή σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Η κυρία Ροδούλα Ζήση από την Ελλάδα έχει το λόγο να χαιρετήσω αυτή τη συνάντηση να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό ε, της ουγγαρίας και να συγχαρώ την ε, ε, ουγγρική προεδρία της ένωσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον πρόεδρο της επιτροπής και να πω ότι αυτή η συνάντηση κύριε πρόεδρε σημαίνει τελικά πάρα πολλά. ακούστηκαν εδώ κάποιες λέξεις όραμα βούληση πολιτική χαρτογράφηση αναγκών δυνατοτήτων ακούστηκαν πραγματικά πολύ σημαντικά ζητήματα που δείχνει τελικά ότι αυτός ο διάλογος επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο πρωθυπουργός της ουγγαρίας ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει ανάγκη και από τη διεύρυνση και από την εμβάθυνση. όμως δεν μπορεί η ένωση ούτε κάποιος από εμά να χειραγωγήσει αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται. η χαρτογράφηση της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να συναντηθεί με την πολιτική ιστορία με το χάρτη της ιστορίας των δυτικών βαλκανίων. πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτές οι χώρες αυτή η περιφέρεια της ευρώπης μπορεί με την ένταξή της στην ευρωπαϊκή ένωση με τον πολυπολιτισμό της με την κουλτούρα και την ιστορία της να δώσει προστιθέμενη αξία στις αξίες της συνολικές που έχει η ευρωπαϊκή ένωση τις αξίες της ειρήνης της αλληλεγγύης του πολιτισμού και της προόδου. είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το όραμα που, έχει ανάγκη ο, ο κόσμος της ευρωπαϊκής ένωσης ο κόσμος των δυτικών βαλκανίων να δει να εφαρμόζεται αυτό το όραμα είναι τα συναισθήματά μας που γεννούν τις σκέψεις μας που είναι τα παιδιά μας και αυτές οι σκέψεις στην πολιτική στην ανάπτυξη στη ζωή μπορούν πραγματικά να πραγματώσουν όνειρα και προσδοκίες. Δεν χρειάζεται όμως να βιάζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες. Είμαστε υπέρ της ενταξιακής πορείας ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά οι χώρες μπορούν να λύσουν διάφορα ζητήματα, όπως τότε. Υπήρχε πάντα μια χάρτα πολυπολιτισμού. Εκεί τότε με τον Ρίγα, τον Βελεστινλή, τον πατριώτη μου, τον πρόγονό μου, που μπόρεσαν οι λαοί αυτοί και υπήρξαν με συνεργασία και με αλληλεγγύη άρα θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες όχι απλά τις ισορροπίες ε, τις πρωτοβουλίες εκείνες που στηρίζουν τις κοινωνικές τις πολιτικές προσπάθειες και προσδοκούν βεβαίως και στηρίζουν αυτό που είπε ο πρόεδρος της επιτροπής την ανάγκη της συνένεσης των πολιτικών κομμάτων μπροστά στο στόχο μπροστά στο όραμα που πρέπει να πραγματοθεί η ελλάδα στηρίζει αυτή την προσπάθεια στηρίζει την ευρωπαϊκή ένωση την ε, ε, ουγγρική προεδρία στηρίζει την επιτροπή σε αυτή την προσπάθεια. άλλωστε η ατζέντα της θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται και με τον οδικό χάρτη που αναδεικνύουμε και προσπαθούμε ξανά να δώσουμε για το. 2014. και πάλι σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο κύριος Λουίς Ροντρίγκες από... Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε του ε, Ουγγρικού Κοινοβουλίου, κύριε ε, Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Μπαρόζο, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την ευκαιρία. Επίσης θέλω να αναφερθώ στην προσωπική εκτίμηση που έχουμε για τον πρέσβη της Ουγγαρίας στην Λισαβόνα. Έκανε εξαιρετική δουλειά ο πρέσβης. Ανέπτυξε εξαιρετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ουγγαρίας και Πορτογαλίας. Και είναι μεγάλο προτέρημα του ότι γνωρίζει η Πορτογαλικά. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή τη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά και για τον ρόλο που προβλέπεται στα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ. Πολλές φορές φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια κατά κάποιο τρόπο αμελούνται ή αγνοούνται. Δεν είναι τόσο σημαντικά πολλές φορές σε αυτή την οικοδόμηση εδώ όμω κάνουμε αυτό το οποίο συνέβη εχθές. Ε, με βεβαιότητα τονίζεται η συμμετοχή, η ε, σημασία της συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνα τα κράτη που θα είναι στο μέλλον μέλη και εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάζοντας το χάρτη της Ευρώπης καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια αναπόφευκτη πορεία. Νωρίτερα ή αργότερα θα γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό. Ακούσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν υπάρχουν ακόμα. Όμως η Ευρώπη έχει μια πορεία που πρέπει να πορευθεί και σε αυτόν τον όλο και πιο περίπλοκο κόσμο. Πέρα από την πολιτική που χαιρετίζω εδώ για τη διεύρυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρθηκε επίσης, έχουμε και την πολιτική της παγίωσης και ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σημαντικό στοιχείο. Σε αυτή την παγίωση με την διεύρυνση είναι στοιχεία που δεν μπορούν να ε, αποσυνδεθούν. Η διεύρυνση είναι πάρα πολύ σημαντική σημαντική για την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουμε την πολυμορφία την πολιτισμική, την πολιτική μας ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εμβάθυνση. Με αυτές τις διαφορές πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη πιο δυνατή. Στην Πορτογαλία δεν είναι, ε, παρότι υπάρχει απόσταση από τα Δυτικά Βαλκάνια γεωγραφική, δεν υπάρχει όμως ε, σε σχέση με την πολιτική κατεύθυνση. Φαίνεται ότι είμαστε απομακρυσμένοι, όμως ε, είμαστε πολύ κοντά. Φαίνεται, η Πορτογαλία πρέπει να βρίσκεται παράλληλα ευθυγραμμισμένη σε αυτές τις προσπάθειες για να συνεισφέρουμε για τη διεύρυνση με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι, να συνεισφέρουμε από πλευρά μα. Διότι έχουμε εμεί εδώ πραγματικά την κοινή δέσμευση. Θέλουμε να συνεισφέρουμε για να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά όλο και περισσότερο και κάθε φορά με μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να δώσω εδώ στα κράτη τα οποία βρίσκονται εδώ παρόντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από πλευρά τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιρτσεφ παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Είμαι βαθιά πεισμένος ότι η ευρωπαϊκή προοπτική ε, και η προοπτική των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να υλοποιηθεί. Οι τριβές και οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν είναι αντιπαραθέσεις και διαφορετικές γνώμες για τον ρυθμό, την ταχύτητα, τις πιθανές πρόσθετες προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν από πλευράς μας για να αποφύγουμε προβλεπόμενα προβλήματα και να αποφύγουμε δυσάρεστε εκπλήξεις. Υπό αυτό το πρίσμα πιστεύω ως προσθήκη σε σχέση με τους πολιτικούς και τους ευρωβουλευτές θα πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες. Στα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να ακούσουμε τις φωνές των διανοουμένων και των ειδικών, των πραγματογνωμόνων. Αυτές οι φωνές πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη, να είναι πιο δυνατές. Δεν είμαι βέβαιος αν τα όσα γίνονται επαρκούν. Είναι μια πολύ περίπλοκη ιστορία, πολύ ιδιόμορφη περιοχή με πολύ ε, ξεχωριστή ιστορία και παραδόσεις. Καμιά φορά βλέπουμε εδώ προβλήματα συμφέροντα συνοριακά, συνασπισμών, ε, διαφορετικά προβλήματα. Πολύ σωστά προαναφέρθηκε από τον κύριο Όρμπαν ότι το καθεστώς των διαφορετικών κρατών ε, υπό ένταξη δεν πρέπει να συγχαίρεται από τη μία σε σχέση με την άλλη χώρα. Αυτά τα οποία αναφέρθηκαν για την Κροατία, το Μαυροβούνιο, ε, τη Βοσνία, το, την, με συγχωρείτε, το Μαυροβούνιο είναι, πρέπει να διαφοροποιούνται σε σχέση με κάθε χώρα. Για το θέμα της ονομασίας ε, της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής, γιατί δεν ε, διαπραγματεύονται ε, πραγματικά με ειλικρίνεια σε μια πραγματική βάση συνεννόησης τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Έχουν υπάρξει πολλές φορές ψηφίσματα, προτρέπουμε και ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, να προχωρήσουν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Όμως αυτό δεν λειτουργεί και δεν προχωρεί. Στην κεντρική Ευρώπη το να αλλάξει μια χώρα το όνομά της. Είναι τόσο δύσκολο να ευρεθεί μια εναλλακτική λύση για το όνομα της Μακεδονίας, λέει ο μιλητής. Αν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη ε, θεωρούν ότι, πρέπει, ότι μπορούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, ας δούμε τι γίνεται με το Κωσυφοπέδιο. Το Κωσυφοπέδιο δεν έχει αναγνωριστεί από πέντε κράτη-μέλη και η πρόοδοση είναι αδύνατη. Πρέπει λοιπόν να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να στα στραφούμε στο βάθος των προβλημάτων και να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο η Μακεδονία, λέει ο μιλητής, ώστε να μπορέσει για παράδειγμα να ε, υπάρξει κάποια αντιμετώπιση σε σχέση με την ε, Σερβία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας ενώνουν και πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην αναζήτηση μιας ε, λύσης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν πολλά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και πρέπει να κάνουν πολλά υπέρ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστούμε την Doris Πάκα για όσα έχει κάνει υπέρ των χωρών αυτών προς την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και έχουμε δύο παρεμβάσεις με γαλάζιες κάρτες. Θα γίνουν τώρα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ωφεληθώ από την παρουσία του Πρωθυπουργού Όρμπαν να του θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύει ότι ο νόμος για την Ουγγρική υπηκότητα αν ωφελεί γενικά την περιοχή και τους διάφορους και τους κατοίκους στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Απάντηση. Ο κύριος Γιάν Μπάουερ μάλλον. Για το Κοινοβούλιο Τσεχικής Δημοκρατίας έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που μου διατίθεται να μιλήσω εκ μέρους της τσεχικής αντιπροσωπείας. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό ο κύριος Ορμπάν και η χώρα του χειρίστηκαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με πολύ επιτυχή τρόπο, πολύ επιδέξιο. Το πιστεύω πραγματικά ε, και είναι ε, σύμπτωση που μιλάμε μετά το Σλοβάκο συνάδελφο, η Ρίστον Παρόδο. Χειριστήκατε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε πολύ δύσκολη εποχή, κύριε Ορμπάν, και η Τσεχική Δημοκρατία αντιμετώπισε πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως η κρίση του φυσικού αερίου Ρωσίας-Ουκρανίας. Εσείς πρέπει να αντιμετώπισετε διάφορα οικονομικά ζητήματα και δεν είσαστε σε καθόλου πιο εύκολη θέση. Και τώρα, αυτό που θέλω να πω, για την περαιτέρω διεύρυνση θέλω να πω κάτι. Άκουσα τις, την ομιλία του Πρωθυπουργού Ορμπάν και του Προέδρου Μπαρόσο και νομίζω ότι περιγράψατε πολύ σωστές θέσεις, περιγράψατε πολύ λογικά το πώς θα έπρεπε να προσεγγίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και είπατε σωστά τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εν λόγω χώρες. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα προς επίλυση και καμιά φορά δεν κάνουμε το σωστό αλλά μόνο αυτό που είναι πολιτικά εφικτό. Ξέρω ότι το θέμα της συζητήσεως δεν είναι η οικονομία αλλά τα Δυτικά Βαλκάνια. Όμως αρκετοί προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι κάποιες αντιπροσωπείες κάποιων σημαντικών κρατών μελών απουσιάζουν από τη συνεδρίαση. Κύριε Πρωθυπουργέ Ορμπάν, κύριε Μπαρόσο, τι πιστεύετε, θεωρείτε τα οικονομικά μέτρα που λάβαμε όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας ή το οικονομικό πακέτο αυτά τα μέτρα είναι σωστά είναι σωστοί οι μηχανισμοί για να ισχυροποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρατήσει τη δύναμή της, θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα και μεταβίαστα θα μπορεί να διευρυνθεί ή να εμβαθυνθεί στο μέλλον. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από το Γκρικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Το 2011 <clears throat> μπορεί να είναι ένα ορόσημο και με ένα σημείο καμπής όσον αφορά τη σταθεροποίηση των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας και ε, λαμβάνοντα υπόψη και την ε, ε, αρνητική τροπή των πραγμάτων. Η συνεχιζόμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί ίσως να τροχοπεδηθεί και να σταματήσει αν η ολοκλήρωση σε σχέση με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων επιβραδυνθεί και κάτι τέτοιο θα είχε πραγματικά ανυπολόγιστες ε, επιπτώσεις. Γι' αυτό προτείνω ότι δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία πραγμάτων. Και λαμβάνοντας υπόψη την ανακυκλούμενη Προεδρία, αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στην ένταξη των Δυτικών Βαρκαλίων. Βαλκανίων. Είναι μια περιοχή ακριβώς στο ε, σταυροδρόμι βορρά-νότου Ανατολής Δύσης. Ακριβώς αυτό είναι, αυτή είναι μια κέρια περιοχή για πολιτισμικά θέματα και πολιτισμική πολυμορφία που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη. Αρκετοί ομιλητές σήμερα προανέφεραν και τόνισαν ότι ο πολιτισμικός διάλογος θα μπορεί να είναι καταλήτης σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Και έτσι θα έπρεπε να δρά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να συνεισφέρει και να συνεχίσει, να συνεχίσει αυτόν τον πολιτισμικό διάλογο υπό την παραδοσιακή συνεργασία που εξελίσσεται και οι εθνοτικές μειονότητες, οι εθνοτικές ομάδες ε, οι ίδιες θα πρέπει επίσης να εμπλέκονται μέσα στο πλαίσιο αυτών των καταλυτικών διεργασιών. Η, ο πολυσχηδής χαρακτήρας πολιτισμικά αυτής της ε, περιοχής ε, μπορεί να ε, εξυπηρετήσει ως πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι ένα υπόδειγμα και τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η Ευρώπη σε ένα καριδότσουφλο, η Ευρώπη σε μικρογραφία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνιστόσα στην ευρωπαϊκή πολυμορφία και αυτή τη συνιστόσα πρέπει να εντάξουμε ολοκληρώνοντας την Ευρώπη. Και θα πρέπει οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες να συνειδητοποιήσουν και να γνωρίζουν ότι έχουν μια θέση που τους αρμόζει, νόμιμη θέση στην μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών. Και σε σχέση με την εξέλιξη αυτή θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους επόμενους μήνες. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε από πλευράς των κρατών μελών να προαγάγουμε τα συμπεράσματα αυτά για να προαθούν οι ε, διαπραγματεύσεις και να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στάντλερ από την Αυστρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρωθυπουργό να τον συγχαρώ διότι η Ουγγρική Προεδρία με εξαιρετικό τρόπο προχωρεί στις δράσεις της και τα καταφέρνει. Στις αρχές της Προεδρίας υπήρξαν κάποιες σημαντικές δυσκολίες, τις οποίες όμως δεν θεωρήσαμε σωστές και ε, δικαιολογημένες αυτές τις δυσκολίες που προκλήθηκαν. Τώρα για τη συζήτηση για τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Υπό την εμπειρία που έχουμε ε, συσσωρεύσει πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα σε σχέση με τις χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η διεύρυνση με τις χώρες αυτές δείχνει όχι υπερβολική ταχύτητα αλλά πρέπει στην σωστή προετοιμασία να βασιστούμε. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει πιο πολύ. Είναι σκόπιμο αυτές οι χώρες να έχουν την προοπτική της ένταξης και την προοπτική της ιδιότητας ε, υποψήφιας χώρας προς ένταξη ως ε, κίνητρο για να λάβουν υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που πρέπει να κάνουν όπως για παράδειγμα η Αλβανία τεράστιες προσπάθειες προσπάθειες που απαιτούνται. Αντίστροφα όμως, εκεί όπου έχει προχωρήσει μια χώρα πολύ, όπως η Κροατία, θα πρέπει χωρίς προβλήματα γοργά να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να ενταχθεί η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι η Κροατία σε σχέση με άλλες χώρες υποψήφιες ή πρώην υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προπολού υλοποιήσει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που θα επέτρεπαν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία παρατήρηση. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λαοί, τα έθνη των Βαλκανίων. Η ιστορική πείρα δείχνει σε σχέση ε, με αυτά τα θέματα ότι μια ιδιαίτερη ευαισθησία απαιτείται. Θα ήθελα να απευθύνω το εξή προ τη συνάδελφο Πακ. Δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση των λαών των Δυτικών Βαλκανίων να του κάνουμε μαθήματα ή κατήχηση ω δάσκαλοι. Πρέπει με ιδιαίτερη ευαισθησία να αντιμετωπίσουμε την πολιτισμική πολυμορφία και τι ταυτότητε ε, των ε, λαών των Βαλκανίων το γνωρίζουμε αυτό από την πείρα μα Και είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη και την ιστορία. ιστορία που είναι πολύ περίπλοκη και πολλέ φορέ δημιουργεί μια αδιαφάνεια λόγω περιπλοκότητα. Και εδώ πρέπει σε σχέση με την Ουγγαρία, με, τις, ε, ιστορική, με την ιστορική πείρα σε σχέση με τα Βαλκάνια, να προχωρήσουμε με ευαισθησία. Ευαισθησία, αλλά να λάβουμε υπόψη και το θέμα τη ονομασία, που για πολλού φαίνεται κάτι το αποξενωμένο ή απόμακρο. Πρέπει να δείξουμε κατανόηση για την ελληνική κοινωνική που ε, για την ονομασία επιβαρύνεται ιστορικά από την ιστορική παράδοση, την ίδια την ιστορία της Ελλάδας. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους δύο αυτούς λαούς ε, διμερώς οι ίδιοι, οι ίδιες αυτές οι χώρες επεξεργαζόμενες ε, το παρελθόν και την παράδοση να αντιμετωπίσουν το θέμα της, ονομασίας. Δεν είναι μόνο η ονομασία, είναι και άλλες παραδόσεις και ιστορικές, ε, ιστορικά κληροδοτήματα. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν έτσι να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Γκαστούσκοβα από την γερουσία της τσεχικής δημοκρατίας. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να δώσω ξανά την προεδρία της, να δώσω την προεδρία της συνεδρίας στον κύριο Μαρτίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Μπαρόσο, κύριε Πρωθυπουργέ Ορμπάν, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούσεκ, και να συγχαρώ και την Ουγγρική Προεδρία για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση. Είναι πολύ χρήσιμη επίση εκδήλωση και για τα κάτι μελη της Ευρωπαϊκής Ενώσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους εκπροσώπους, ελπίζω, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ακούσαμε ομιλίες που αναφέρθηκαν στο ρόλο της παιδείας και του πολιτισμού, αναφέρθηκαν στην κοινή ιστορία που δεν θα πρέπει να μας διαιρεί, να μην διαιρεί κυρίως τους νέους, πρέπει η ιστορία να τους ενώνει, αντίθετα. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί, αλλά το όλο εγχείρημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που έχει σημεύσει σαν παράδειγμα. Θυμηθούμε τα λόγια του Ρομπέρ Σουμά, που ήταν Ευρωπαίο πολιτικό και είχε ένα όραμα για μια ολοκληρωμένη Ευρώπη και το είχε το όραμα αυτό και έγραψε γι' αυτό στη φυλακή και έδωσε στο ευρωπαϊκό αυτό εγχείρημα την αναγκαία δύναμη έδωσε σαν και στο όραμά του για συμφιλίωση, για συγνώμη και ας μην και πόσο ισχυροί είμαστε όσον αφορά τον οικονομικό τομέα σαν Ενωμένη Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σημαντική προοπτική για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και για μας όμως. Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας όσο μεγάλα και αν είναι αυτά αν κινηθούμε ενωμένοι. Σας διαβεβαιώ ότι η τσεχική δημοκρατία σίγουρα θεωρεί τη διεύρυνση σαν σημαντική διαδικασία ανεξάρτητα από το κατά εάν μιλάει κανείς σε εκπρόσωπο της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης αυτών των χωρών. Ε, ε, ε, θέλω να είναι επιτυχής οι διαπραγματεύσεις και έχουμε καλή τύχη και για αυτό το θέμα και για άλλα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε σε σχέση με την Προεδρία που ανέλαβα θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που καταβάλει το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και για να υπάρξει η ε, βοήθεια και υποστήριξη και σίγουρα και με την παρουσία τόσων υπαλλήλων και ιδιαίτερα από πλευρά σας την αδέρφου Πέρτσικ, Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για ε, τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και τώρα θα λάβει τον λόγο στη συνέχεια για να συνεχίσουμε με αυτή τη συζήτηση ο γερουσιαστής Ερνάντεθ από την Ισπανία παρακαλώ σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη Ισπανικής Αντιπροσωπείας τη Γερουσία της χώρας μας θέλω να καταδείξω τη δέσμευση τη Ισπανία για την ευρωπαϊκή προ... προοπτική των Βαλκανίων και να πω ότι είναι πάντα σταθερή και σαφή αυτή η προοπτική όπω και κατά τη διάρκεια τη δική μα προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προώθησε η Ισπανία την ε, συνάντηση σε υψηλό επίπεδο στο Σαράγεβο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μεταξύ όλων των χωρών χωρών της Ζώνης και της Ένωσης. Θέλουμε να συνεχιστεί η αναζήτηση λύσης μεταξύ των αρχών της Ελλάδας και της ε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της ε, Μακεδονίας για το επίσημο όνομα αυτής της χώρας, την ονομασία που θα δώσει την δυνατότητα να προχωρήσει με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξή της αυτή η χώρα υστερότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν επιληθεί αυτό το ε, επίμαχο σημείο. <clears throat> θα πρέπει να υπάρξει προώθηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. ολοκληρώθηκε ε, η, ε, το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίων, το θέμα της ιδιότητας υποψήφιας χώρας στο Μαυροβούνιο, καθώς επίσης και η Συμφωνία Σταθερότητας, ε, Σταθεροποίησης και εταιρική σχέση με τη Σερβία. Και έτσι το 2011 μπορεί να είναι ένα νέο έτος, όπως μπορεί να καταδείξει αυτή η συνάντησή μας εδώ που έχει συγκληθεί μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία πρόοδος που θα σημειωθεί για τις χώρες αυτές με την έγκριση ε, για την Αλβανία και τη Σερβία χωρών υποψηφίων προς ένταξης. Ε, και η αντιπροσωπεία της Ισπανίας παραδοσιακά ήταν πάντα υπέρ της διαδικασίας ε, σταθεροποίησης και εταιρική σχέσης και της ένταξης ως προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτή την προοπτική και εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη αυτού του ευκταίου στόχου. Και από πλευρά μα, εξ ονόματο τη Γερουσία τη Ισπανία, θέλω να ευχαριστήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Τώρα θα λάβει τον λόγο ω τελευταίος αγορητη ο κύριος Οπρέα τη της Ρουμανικής Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω εδώ μια κάποια αμηχανία. Αμηχανία πρέπει να πω για την έναρξη αυτής της συζήτησης, αυτής της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ενός ε, βουλευτή από την Ρουμανία και μιας εκπροσώπου της Αλβανίας. Είναι ένα τυπικό παράδειγμα θα έλεγα των εντάσεων που εμφανίζονται, ε, αναφύονται στα Βαλκάνια αυτή η περίπτωση. Όμως πιστεύω ότι δεν αντανακλά σε καμιά περίπτωση μια εχθρότητα, μια εθνική, εθνοτική εχθρότητα. Πολλά πράγματα μας συνενώνουν και πιστεύω ότι η φιλία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των Αλβανών και των Ρουμάνων δεν μπορεί να υποστεί αρνητική επίπτωση από τέτοιου είδους ανταλλαγές απόψεων. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ε, υπήρξε συνεργασία και για την ε, δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου στα Βαλκάνια από πλευράς μας και ένα δίκτυο που με κανένα τρόπο, καμιά πολιτική εχθρότητα δεν θα μπορέσει να καταστρέψει. Και εδώ ακριβώς ε, οι νέοι είναι εκείνοι που θα πετύχουν, όχι οι πολιτικοί μόνο, αλλά οι νέοι κυρίως ώστε η Ευρώπη να βασίζεται, να έχει στη διάθεσή της μια απόλυτη τέλεια ολοκλήρωση σε σχέση με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, ολοκλήρωση που θα επιτύχει. Αυτό είναι ευταίο ώστε όλη η πολιτισμική πολυμορφία να αντανακλάται των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι και ο τελικό στόχο που πρέπει να ευδοκιμήσει. Με όλε αυτέ τι επιτυχίε που αναμένουν και πρέπει να επιτελεστούν στο μέλλον, στο άμεσο απότερο μέλλον πρέπει η παιδεία εκπαίδευση στα σχολεία να διαδραματίσει η παιδεία και η εκπαίδευση ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας Έλληνας ε, για παράδειγμα ε, σε σχέση με έναν, με έναν εκπρόσωπο των, ε, της Μολδόβας αναφέρθηκε αυτή η πτυχή ακριβώς αυτής της σημαντικής συνεισφοράς για τα Βαλκάνια μιας περιοχής που είναι ζώνη υψηλών πιέσεων και εντάσεων αλλά και όμως πραγματικά θα έλεγα ιδιαίτερα σε βάθος προσέγγισης χρειάζεται αυτή η ενδυνάμωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο να ενδυναμωθεί αυτή η προοπτική πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια ζώνη ιδιαίτερα αξιόλογη, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρέπει να κάνουμε πολλά για αυτού. Και εμεί του χρειαζόμαστε, δεν είναι μόνο εκείνοι που μα χρειάζονται. Χρειαζόμαστε ο ένα τον άλλον αμοιβαία. Αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται εδώ γύρω στον αγοριτών που είχε καθοριστεί ως κατάλογος για αυτό το γύρο. Ευχαριστούμε όλους για τις παρεμβάσεις, τις ιδέες τις προτάσεις τους. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος ε, Ντουράν Μπαρόζο και ο κύριος Πρωθυπουργό Όρμπαν. Στο σημείωμα που μου προετοίμασαν εδώ μου λένε ότι σύντομε λέει παρεμβάσει, διότι ήθιστε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχουν απαντήσει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου πιέζει όμως ο χρόνος βασιζόμαστε στην ε, ε, θα έλεγα κατανόηση των αγορητών και έτσι δεν πρόκειται να αφαιρεθεί το μικρόφωνο αλλά παρακαλώ πλήρως ελεύθερα να μπορέσετε να παρέμβετε στις οικοδομητικές, επικοδομητικές αυτές παρεμβάσεις. Πρώτα λοιπόν θα λάβει τον λόγο ο κύριος Μπαρόζο μου έχουν σημειώσει εδώ. Κύριε Ντούρα Μπαρόζο έχετε τον λόγο παρακαλώ θα σας ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Um, so uh, σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση και να απαντήσω συγκεκριμένα συγκεκριμένες ερωτήσεις που μου απευθύνθηκαν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον διορισμό του πρεσβευτή μας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Χθες η Βαρόνη Άστον μας ενημέρωσε λέγοντας ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία της επιλογής έψαχνε να βρει μια μεγάλη προσωπικότητα επιφανή διπλωμάτη γιατί θέλουμε να είναι ισχυρή η εκπροσώπησή μας. Διότι η νέα αντιπροσωπεία μας, η πρεσβεία μας εκεί, θα έχει τη, σωσ... συνηθισμένη δουλειά μιας αντιπροσωπείας, αλλά και το ρόλο ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα πολιτικά ζητήματα εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής από την κυρία, από τη Λέδη Άστον. Όσον αφορά το ερώτημα που μου ετέθη, για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και τα μέσα τα διαθέσιμα. Ελήφθησαν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, που μπορούσαμε να λάβουμε, είναι φιλόδοξα, εγώ θα προτιμούσα να πηγαίναμε ακόμα πιο πέρα. Σε συντονισμό οικονομικών πολιτικών, όλα αυτά η συνένεση ήταν πολύ καλή αυτή που επετεύχθη στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε περισσότερα εργαλεία τώρα, είναι σημαντικά τα εργαλεία, αλλά δεν τα πάντα. Πολύ συχνά στην Ευρώπη αναφερόμαστε πολύ συχνά σε θεσμού και διαδικασίε και λησμονούμε στην πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα και προθυμία συνεργασία. Αν οι κυβερνήσει τώρα πάρουν τι αποφάσει όσον αφορά την οικονομική ενοποίηση, δια, διαθωτικέ αλλαγέ και μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα σε συνεργάσιμο πνεύμα με τα παρόντα εργαλεία, τα παρόντα μέσα και με σεβασμό ε, του ρόλου των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο. Το πιο σε ερώτημα ήταν του Λόρδου Evans. Αφορούσε το πώς να εμπλέξουμε εκείνα τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται λιγότερο για την ε, διεύρυνση. Πώς να τα κάνουμε ενδιαφερθούν. Πράγματι το ενδιαφέρον όσον αφορά τη διεύρυνση, να το πούμε, είναι διαφοροποιημένο στα διάφορα κράτη-μέλη και στα κράτη-μέλη διάφορα, διάφορα τμήματα τη κοινή γνώμη έχουν διαφορετική άποψη. Κάποιο αναφέρθηκε στην κόποση από τη διεύρυνση. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ξεκαθαρίσω, δεν έχουμε κόποση όσον αφορά τη διεύρυνση. Πάντα είμαστε αφοσιωμένοι στη διεύρυνση. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρισίμου σημασία για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είπα στην αρχή τη δήλωσή μου ότι η ευρωπαϊκή διεύρυνση δεν ήταν μόνο μία από τις επιτυχέστερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την πρόθεση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της σχεδόν ανοιχτών οικονομιών και την επικράτηση του κράτους δικαίου αλλά πιστεύω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία αν το δούμε από τη σωστή προπτική. Αν βάλουμε σε προπτική από τη διεύρυνση από τα 6, πρώτα 9 μέλη, στα 27 τα σημερινά μέλη και σύντομα κι άλλα, είναι κάτι φανταστικό αν σκεφτεί κανείς τι αντιπροσωπεύει. Αυτή η δημιουργία της ενότητας μετά τα φοβερά γεγονότα του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που ε, συνέβη στην Ήπειρό μας. Το θαυμάζω αυτό και σας μεταφέρω αυτό το θαυμασμό. Όταν συναντούσα Αμερικανούς, οι Κινέζους, οι Ρώσους φίλους μας ή άλλους εταίρους, ένα από τα θέματα που θαυμάζουν περισσότερο για την Ευρώπη είναι αυτό. Πώς καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, να πετύχουμε αυτή τη διεύρυνση. Έχω βαθιά συναισθήματα για την διαδικασία τη διεύρυνση. Αυτή είναι η θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και σαφεί. Δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τα πρότυπα, τι προδιαγραφέ. Οπότε πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στι υποψήφιε χώρε και στι χώρε που θέλουν να γίνουν υποψήφιε χώρε. να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουν και αυτέ τη δουλειά του. Και δεν νομίζω ότι βοηθούμε κανέναν όταν προσπαθούμε να πούμε ότι από εμά εξαρτάται την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τι χώρε. Κανεί δεν αντικαθιστά τι ίδιε τι χώρε να επιλύσουν τα προβλήματά του. Όσον αφορά τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει, όσον αφορά το κράτο δικαίου, όσον αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορά, όσον αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητηθεί ειλικρινά. Ε, νομίζω ότι έγινε ειλικρινή συζήτηση. Πώ τώρα να ε, προσελκύσουμε και του άλλους συμμετάσχουμε, ακριβώς αυτό που κάνουμε, συμμινομιλώντας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο Λουί Ροντρίγκο, από την Assembleia de República τη Πορτογαλία, είπε, από τη συνέντευξη στην Πορτογαλική, ότι η Πορτογαλία υποστηρίζει την ευρωπαϊκή διεύρυνση προ τα Δυτικά Βαλκάνια και νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό το μήνυμα. Δεν είναι μόνο οι χώρε που είναι πιο κοντά στα Δυτικά Βαλκάνια που έχουν αυτή τη στάση, αλλά και χώρες που δεν είναι τόσο κοντά καταλαβαίνουν πολιτικώς πώς, πόσο σημαντικό είναι αυτό, ούτω ώστε ε, να δούμε ότι η επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντική. Στην αρχή της δεύτερης θητείας μου πήγα σε αυτή την περιοχή για να τους δείξω ακριβώς πόσο σημαντική είναι η διεύρυνση. Και τώρα διεξάγεται και αυτή η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι η προσχώρηση της Κροατίας που ελπίζω να γίνει σύντομα, είμαστε στην τελευταία φάση διαπραγματεύσεων, ελπίζω να είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτός να ρίξουμε κάποιο φως, να εστιαστούμε στη διεύρυνση. Ελπίζουμε να ξεκινήσει μια σημαντική συζήτηση πάνω σε αυτό στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαι ειλικρινής, ε, καμιά φορά απογοητεύομαι διότι κράτη-μέλη που, που κερδίζουν τόσο πολλά από τη διεύρυνση Τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν εξηγούν ειλικρινά πόσο σημαντική είναι η διεύρυνση όχι μόνο για τα κράτη που γίνονται μέλη, τα καινούρια κράτη, αλλά και για τα παλιά κράτη-μέλη. Μεγάλη αύξηση του εμπορίου. Τι σημαίνει αυτό για την ενιαία αγορά. Η ανάπτυξη του εμπορίου λοιπόν, η, ανάπτυξη, η αύξηση των ωφελών για τα πρώην ε, κράτη-μέλη της παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι πολύ σημαντικά το ωφέλη με τι και αυτό δεν ακοινώνεται στον τύπο, στα μέσα ενημέρωση και στο κοινό. Και έτσι δυσκολεύονται οι εθνικοί πολιτικοί να πούν θέλουμε να προχωρήσουμε με τη διεύρυνση. Διότι σε εποχές οικονομικής κρίσης οι πολίτες βέβαια ανησυχούν. Φυσικό είναι σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης οι άνθρωποι να γίνονται πιο αμυντικοί. Αν οι ηγέτες σε εθνικό επίπεδο δεν εξηγούν πόσο σημαντική είναι η διεύρυνση, τότε βέβαια δεν πρέπει να περιμένουν και μεγάλο ενθουσιασμό από τους πολίτες. Γι' αυτό πραγματικά χρειαζόμαστε μια συζήτηση όσον αφορά τη διεύρυνση, τα ωφέλη της διεύρυνσης, τι σημαίνει πολιτικά, τι σημαίνει οικονομικά ε, για την Ένωσή μας. Και νομίζω ότι οι συνεδριάσεις όπως αυτή η σημερινή πραγματικά είναι σημαντικές. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε νομίζω, ο κ. Μποστινάρου νομίζω τέθεσε. Αυτό είναι ο ρόλος των πολιτικών οικογενειών, των πολιτικών κομμάτων. Και εφόσον είμαι εδώ και μιλώ σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να το πω και αυτό, να το ξεκαθαρίσω. Στα Βαλκάνια και σε άλλε επαφέ που έχω, τι βλέπω, ότι καμιά φορά κάποιε από τι πολιτικέ δυνάμει αμφισβητούν την νομιμότητα του Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να είμαστε ειλικρινεί γι' αυτό. άλλο, εγώ είμαι πολιτικός, ήμουν πρωθυπουργό στη χώρα μου, ηγέτης αντιπολίτευσης, μου αρέσει η συζήτηση πολιτική. Άλλο αυτό. Να, να πηγαίνουμε σε μια χώρα. Και όταν η ηγέτης αντιπολίτευσης μας λέει ότι η κυβέρνηση δεν είναι νόμιμη, δεν σέβεται την ελευθεροτυπία και η κυβέρνηση λέει ότι η αντιπολίτευση δεν είναι σωστή όσον αφορά, σαν αντιπολίτευση όσον αφορά τα δημοκρατικά πλαίσια, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν θέλουμε και αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσεί τα μέλη του Εθνικού Εθνικών Κοινοβουλίων θέλετε να υποστηρίξετε τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, ένα πράγμα που σας συστήνω να κάνετε θερμά είναι να αυξήσετε τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ πολιτικών οικογενειών στα κοινοβούλια σας για να δημιουργήσουμε, πώς να το πω, ένα, μια δημοκρατική νοοτροπία, περισσότερο δημοκρατική νοοτροπία και σχέσεις μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Ζωηρή συζήτηση αλλά σταθερή δημοκρατία. Χρειάζεται να προωθηθεί αυτή η κουλτούρα της συνένεσης και του συμβιβασμού. Όχι να μειωθεί η δημοκρατική συζήτηση και η ζωηρή συζήτηση που γίνεται σε όλες τις δημοκρατίες μας, αλλά για να προωθήσουμε ε, αυτού του είδους την ενοποίηση, παγίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντική αποστολή και για σας και για μας σαν πολιτικούς. Όπω είπα και πριν, η διεύρυνση δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, δεν είναι τεχνοκρατική διαδικασία. Χρειαζόμαστε κινητοποίηση των κοινωνιών, είναι μια μεταμόρφωση ε, για να ανοίξουν οι κοινωνίε, για να ανοίξουν ε, οι οικονομίε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και κατά την άποψή μα, αυτό που θα κάνουμε εμεί, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνουμε τα πάντα για να κρατάμε επίκαιρο το θέμα. Ευχαριστώ ειλικρινά την Ουγγρική Προεδρία και τον Πρωθυπουργό Ορμπάν για την αποσύρωσή του για αυτό το θέμα. Και φέτο, όπω και πέρσι, το φέτος και το φετινό έτο μπορεί να είναι ε, ένα έτο πρόοδου για τη διεύθυνση Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το είπα όταν επισκέφθηκα τα Βαλκάνια, θα το επαναλάβω και τώρα στην επίσκεψη που θα κάνω τον επόμενο μήνα. Υπό την προπόθεση βέβαια ότι αυτέ οι χώρε αποφασιστικά θα ακολουθήσουν το δρόμο των μεταρρυθμίσεων του ώστε να μπορούν να γίνουν όχι μόνο μέλη τη ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι ήδη, αλλά πλήρη μέλη τη Ένωσή μα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, για όλου μα. Είσαστε πάντοτε πηγή έμπνευση εσείς και αυτά τα οποία λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική διαπαιδαγώγηση την οποία έχετε αναλάβει να μεταλαμπαδεύσετε και όλοι μας επομένως ωφελούμεθα από αυτό και τώρα να δώσουμε τον λόγο με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση Ε, στην ε, Ουγγρική Προεδρία ε, για, για επίσης οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πόσο εύστοχα κρατά το πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φίλο Βίκτορ Όρμπαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θέλω να σας απαντήσω σε κάτι το οποίο αφορά τη χώρα μου την Ουγγαρία. Μίλουμε για το θέμα της ε, ηθαγένειας που απονέμεται εις τους Ούγγρους που κατοικούν εκτός της χώρας, τους Ούγγρους της Διασποράς. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις δυσμενείς διακρίσεις που σοβούν σε κάποιες γειτονικές χώρες, σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε το θέμα της διπλής ηθαγενείας. Στην Κροατία αυτό είναι σύνομο. Στη Σερβία και στη Ρουμανία επίσης. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ότι η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να έχει την δυνατότητα απονομής δεύτερης, διπλής ηθαγένεια και εν πάση περιπτώσει έτσι θα έρθει και αυτή η δυσμενή διάκριση. Τώρα, να σας πω για κάποια θέματα της ε, Ουγγρική προεδρία, ευχαριστώντα σα για τα καλά σα λόγια. Βεβαίω, ακόμα έχουμε μπροστά μας δρόμο, επομένως θα μπορούσα να πω ότι είναι κάπως ε, πρόωρα τα συγχαρητήρια γιατί μπορεί να και τελικά να αποτύχουμε. Πάντως ξεκινώ με μια γενική παρατήρηση. Όταν αρχίσαμε την πορεία της Προεδρίας λάβαμε μια στρατηγική απόφαση. Είπαμε να δούμε κατά πόσο είναι η Προεδρία θα είναι ένα φεστιβάλ, ένα πάρτι, ένα διαγωνισμό ομορφιά ή θα είναι 6 μέρε σκληρή δουλειά. Αυτό το τελευταίο διαλέξαμε και έτσι χαράξαμε την πορεία τη Προεδρία και είπαμε θα πάει ψηλά ο πύχη για την οικονομική διακυβέρνηση. Θα δούμε τι θα γίνει με την ενεργική πολιτική, να δούμε τι θα γίνει με του συγκάντου, να δούμε τι θα γίνει ε, με τη διεύρυνση. Αυτά αυτοί είναι οι βασικοί άξονε που χαράξαμε ότι θα μα απασχολήσουν. Τέτοια ρότα αποφασίσαμε να πάρουμε και επομένω Ελπίζουμε ότι θα έχει σημειωθεί πρόοδος ε, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μας, οπότε και τότε θα αξίζουμε τα ευγενή σας συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά την σημερινή συζήτηση, θέλουμε ο διάλογος με τους εκπροσώπους των κρατών των Βαλκανίων να είναι ειλικρινής και εμείς διατυπώσαμε το τι πρεσβεύουμε με διπλωματικό, με ευγενικό τρόπο, όμως δεν θα πρέπει να παρεξηγείται η στάση μας. Είστε χώρες υποψήφιες για προσχώρηση. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχουν ε, απεσιοδοξίες, επιφυλάξεις, φόβοι και θα πρέπει να προσέξουμε μην παραξενθεί αυτή η κατάσταση. Διότι ξέρετε πριν και εμείς προσχωρήσουμε υπήρχαν επιφυλάξεις και φόβοι πολύ χειρότερα από ό,τι για τη δική σας περίπτωση. Δεν θέλω να δραματοποιήσω την κατάσταση. Είναι δραματική, δεν χρειάζεται να δραματοποιώ περισσότερο και θα πρέπει παρόλα αυτά να μπει στην ατζέντα, στην μοίρα σε διάλεξη το θέμα τη διεύρυνση. Ιδάλω θα περάσουν δεκαετίες και θα είμαστε ακόμα στην κατάσταση. σε τέτοιες διασκέψεις όπως η σημερινή. Θα πρέπει όλα αυτά να τα διεξερχόμεθα. Και θα πρέπει επομένω όλους να τους ευχαριστήσω που συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση. Λέμε ότι τα σύνορα πάνε προς Ανατολάς. Έτσι λέγανε τότε που εμείς προσχωρήσαμε. Έχουμε τα σύνορα της Ελλάδας, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι τα Βαλκάνια δεν είναι πιο ανατολικά από την Ελλάδα. Είναι ένας θύλακας. Άρα έτσι ω τέτοιο θύλακα που είναι μέσα στην Ευρώπη θα τα αγκαλιάσουμε τα Βαλκάνια. Δεν θα βγάλουμε τα σύνορα πιο πέρα. Ήδη κάτι που είναι ευρωπαϊκό θα το αγκαλιάσουμε, να το κάνουμε μέλος της Ένωσης. Άρα, επιφυλάξεις αμφιβολίες, σκεπτικισμός. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα τα διασκεδάσουμε. Πώς με συντονισμένες ενέργειες που ήδη έχουμε αναλάβει. Σύμμαχοι και φίλοι είναι πάρα πολύ βασικό και ε, σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αποδειθεί. Πώς θα κερδίσουμε σύμμαχους και φίλους για αυτή την προσπάθεια. Επομένω, ε, στις διαπραγματεύσεις δικές μας ήμουν πρωθυπουργός, ξέρετε, στο τέλη της δεκαετίας του 90. Και τότε καταλάβουμε ότι ο πιο στέρεος φίλος μας, σύμμαχος, συμπαραστάτης, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ήταν και παραμένει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Φάνηκε από τις αντιδράσεις, από τις απαντήσεις πώς όλα αυτά εκτιμώνται τα οποία αναφέρθηκαν τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της ε, διάσκεψής μας Οι συμπρόεδροι πρέπει να προβούμε σε κάποια σύνθεση των όσων συζητήθηκαν, των όσων αναφέρθηκαν οπότε και με μεγάλη χαρά θα δώσω τις σκητάλη στον συνάδελφο Λάσλο Κόβερ για να αρχίσει αυτή την ε, ε, σύνθεση των όσων ελέγχθησαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφοι. Δεν είναι εύκολο να λαμβάνει στο λόγο μετά τον Όρμπαν, μετά τον Μπαρόζο και να προσθέτει κάτι γιατί τα έχουν καλύψει όλα σε σχέση με όσα συζητήσαμε αυτό το δήμερο. Όμως πρέπει να κάνουμε μια σύνθεση των όσων ακούσαμε αυτό το δήμερο το δήμερο που ήταν τόσο ενδιαφέρον για μένα, διότι άκουσα και χθε και σήμερα τι εισηγήσεις σας που έκαναν τη διάσκεψη πάρα πολύ παραγωγική. Πώς θα πλησιάσουν από πολλές πλευρέ, σε πολλά επίπεδα, τα τρία Βαλκάνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλους τους αγορητές χθεσινούς και σημερινούς. Όλα όσα είπαν νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολλές προσπαθίες μας. Μετά το διήμερο αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχει το τοπίο ξεκαθαριστεί περισσότερο για τις προκλήσεις που αφορούν Ευρωπαϊκή Ένωση και Δυτικά Βαλκάνια. Κατόπιν των όσων ακούστηκαν είδαμε ότι σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπενχάγης τα ζητήματα των μειονοτήτων θα πρέπει πριν την προσχώρηση να έχουν επιληθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για αυτή την ε, περιοχή της Ευρώπης. Επίσης έχουμε τα θέματα δικαιοσύνης, τα θέματα μετανάστευσης. Εκεί θα πρέπει να γίνουν γενναίες μεταρρυθμίσεις. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε επίσης αναβάθμιση των σχετικών ελέγχων. Τώρα όσον αφορά τους πολίτες. Ακούστηκε και διατυπώθηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν και τα φυσικά πρόσωπα, οι πολίτες των χωρών αυτών στην διαδικασία αυτή όπως ακριβώς και τα κράτη. Χρειάζονται κάποια πολιτικά κριτήρια, χρειάζεται παιδεία, να δούμε πώς οι φοιτητέ από τα δυστικά Βαλκάνια θα μπορούν να σπουδάσουν στη Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως και θα πρέπει να παραμείνει η πολιτική πολυμορφία, αλλά θα πρέπει να δούμε και την κοινωνική πτυχή. Να υπάρχει δουλειά. Και έτσι ο κόσμος αυτές τις χώρες να υλοποιήσει τη στρατηγική της Ρώμης. Προσπάθειες λοιπόν από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και ο Πρωθυπουργό Όρμπαν. Σε αυτή τη σύνθεση κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι όλοι, όλοι ετώνησαν πόσο σημαντική υπόθεση είναι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Όλοι επομένως συγκλίνουν στο να διαπιστώσουν ότι υπάρχει η κόποση της διεύρυνσης, όπως επίσης και η κόποση της αναμονής για την προσχώρηση. Παράλληλα φαινόμενα τα οποία θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη διαδικασία της διεύρυνσης. Πολλοί είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη όθηση στα πράγματα. Και ο Πρωθυπουργό Όρμπαν το είπε στην εισήγησή του. Ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία το συντομότερο δυνατόν. Και τι ούτω τρόπος να βοηθήσουμε τις προσπάθειες έμεσα και των άλλων χωρών και σας ευχαριστώ όλους για τόσο είπατε αυτό το διήμερο. Τονίζω και πάλι αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός Όρμπαν. χώρες περιμένουν να γίνουν υποψήφιες, χώρες περιμένουν την προσχώρηση. Για αυτέ όλες τις χώρες ο σημαντικότερο σύμμαχος είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ, σε αυτό το χώρο, βρισκόμαστε και έχω να σα πω ότι έχετε σύμμαχο στις προσπάθειές σας και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση για να καλύψουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και για την προσοχή σας να με ακούσατε. Ο Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε Κεβέρ. Όχι, δεν πρόκειται να επαναλάβω όσα προείπατε. Συμφωνώ με όσα μας αναφέρατε. Θα προσπαθήσω να σε τα συμπληρώσω με τις σκέψεις μου. για όσα άκουσα και από τον πρόεδρο Μπούζεκ να σας πω επίσης ε, το απόσταγμα της δικής μου εμπειρίας για όσα λέμε τα λέμε υπό τις δύο ιδιωτητές μου πρώτα πρώτα ασχολούμαι με τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης όμως εργάζομαι και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψηφίων χωρών. Και μιλώ και για τις υποψήφιες για τις χώρε και για τις υποψήφιες για υποψηφιότητα. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ευρεία αντίληψη, ούτως ώστε να προχωρήσουμε προς αυτή την ενοποίηση της Υπήρου. Φάνηκε μέσα από την εκδήλωσή μας, όπως είπε και ο κύριος Καβέρ, το ότι τέτοιες συναντήσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Έτσι έχουμε επικοινωνία εθνικού, εθνικών και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Όλοι αποκομίζουμε κάτι. Όλοι μαζί προχωρούμε όσον αφορά αυτή την διαδικασία. Αυτή είναι που καλούμεθα να επιτελέσουμε. Όλα αυτά έχουν την νομική τους βάση στη νέα μας συνθήκη της Λισαβόνας. Αντλούμε την νομιμότητά μας και την νομιμοποίησή μας από τους λαούς μας. Οφείλουμε δε να δουλεύουμε για την πρόοδο αυτών των λαών. Συγκεκριμένα τώρα, όσον αφορά τις χώρες αυτές και τα κοινοβουλιά τους θέλω να σταθώ στο εξής. Η συζήτησή μας έρχεται την κατάλληλη ώρα. Η όθηση για να γίνουν τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων πλήρη μέλη των, των δυνατών είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, το χρειαζόμαστε. Όλοι. Και το χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Είναι φανερό ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πλειοψηφία των μελών είναι υπέρ της διεύρυνσης. Δεν θα πρέπει όμως να παρελκύεται αυτή η διαδικασία, διότι έτσι έχουμε κάποιο είδους σπατάλι, φύρα. Είναι μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη. Έχουμε κάποιες δυνάμεις που δεν είναι απλώς ευρωσκεπτικιστές, είναι εχθροί του ευρωπαϊσμού. Και όλοι αυτοί βάζουν τροχοπέδες σε αυτή τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι, η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα υπηρετεί στα συμφέροντα βεβαίως των χωρών εκείνων. Όμως, είναι και για μας τους υπόλοιπους κάτι απαραίτητο. Για όλους που έχουμε πλέον πιστέψει ακράδαντα ότι στην διεθνή σημερινή συγκυρία ή όλοι μαζί θα προχωρήσουμε και θα τα πάμε καλά ή διασπασμένοι θα βυθιστούμε. Και δεν μιλώ μόνο για τις υποψήφιες χώρες, για τις υποψήφιες υποψηφιότητα. Δεν τα λέω μόνο. Αυτά σε επίπεδο θεωρητικό ακαδημαϊκό σας το λέω από την εμπειρία που νιώσαμε στο πετσί μας. Και ο κ. Μπαρόσο και εγώ ίδιος. Ήμασταν και εμεί υποψήφοι για υποψηφιότητα, υποψήφοι για ένταξη. Και πολλέ φορέ αισθανθήκαμε αγανάκτηση γιατί εμεί, οι δικοί μα λαοί που είναι τόσο σημαντικοί ε, στην ιστορία τη Ευρώπη, γιατί, γιατί, γιατί, για κάποιε αιτίε πολιτικέ άσχετε από του λαού μα, μπήκαμε στο περιθώριο. Και έτσι δεν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στην ευημερία που πέρασαν οι υπόλοιπε ε, χώρε που είχαν μπει προηγουμένω. Και το ίδιο ισχύει και για τι 10 χώρε που εντάχθηκαν από την Ανατολική, Δυτική, και Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη που ήταν μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και μετά από αυτή τη διαδικασία μπόρεσαν επομένως να μετάσχουν σε αυτήν την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευημερίας. Επομένως, οι λαοί και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να γίνουν κοινωνία αυτού του οράματος, του υπέροχου. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι και θέμα επανόρθωσης ιστορικής που η ιστορία είχε βάλει στο περιθώριο αυτά τα κράτη, αυτούς τους λαούς φυσικά και πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει κανείς για να κάνει μια διαδρομή να πληρώσει το εισιτήριο. Όμως δεν θα πρέπει ούτε μια δεκάρα να πληρώσουν παραπάνω από όσο πληρώσαμε εμείς για να μπορέσουμε να επιβούμε αυτό το τρένο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Ε, κατακλείδη κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να θυμηθούμε το ότι οι περισσότεροι από όσους μίλησαν και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσον αφορά επίσης τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων πόσο τόνισαν το ότι πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Να μην έχουμε προφάσεις, μην έχουμε δικαιολογίες, να μην υπάρχει τίποτα που να στηρίζει κανένας είδους καθυστέρηση. Να, η Κροατία είναι επιθύρες. Εμείς εμεί από πλευρά μα θα πρέπει, Ζωζέ Μανουέλ, εμεί που νιώσαμε στο πετσί μα τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η καθυστέρηση. Εμεί υποφέραμε την καθυστέρηση. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε την πόρτα του τρένου σε αυτόν που πάει να ανέβει. Άρα, να πούμε ότι η πίτα θα μοιραστεί σε λιγότερους. Όσο πιο πολλοί μετέχουν, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πίτα. Και θέλω να κλείσω αναφέροντας ότι υπό την σημερινή συγκυρία με την παγκοσμιότητα, την οικονομική, την πολυμερή διαχείριση των όσων γίνονται στη διεθνή κοινότητα, καμιά χώρα, κανένα κράτος από μόνο του δεν μπορεί να γίνει παίκτης, συντελεστής στην παγκόσμια σκακέρα μόνο με την ενότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να επηρεάσουμε το γίγνεσθε και να επερμηθούμε των ε, συμφερόντων των Ευρωπαίων και της Ευρώπης και έτσι να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στη διεθνή σκηνή, στην κοινότητα αυτές τις αξίες τις αξίες που χαρακτηρίζουν και οφείλουν να χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή υπόθεση. Ευχαριστώ Ζωζέ Μανουέλ, ευχαριστώ Βίκτορ για τη βοήθειά σας και ευχαριστώ και όλους όσοι έλαβαν μέρος και βοήθησαν. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου που βοήθησαν και εκείνοι που από αυτά τα κλουβιά με τα ακουστικά, όλο ένα και περισσότερο γίνονται, μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε βέβαια και τους τεχνικούς. και στην επόμενη συνάντησή μας που θα γίνει κατά την Πολωνική Προεδρία και ήδη έχουμε ορίσει την ημερομηνία αλλά ακόμα δεν έχουμε ορίσει τη θεματολογία. Κάποια στιγμή το Δεκέμβριο φέτος θα γίνει. Ελπίζω λοιπόν να είναι το ίδιο θετική η εμπειρία όπως είναι και σημερινή. Α, τι για και κάτι τελευταίο, κάτι, μια προσωπική νότα γιατί ορισμένοι από εσά μιλήσατε για το τι παιδεία πρέπει να δώσουμε στους νέους. Καλωσορίζουμε το ακροατήριο όμως που είναι ε, η καλεσμένη δική μου από την Καστίγια Λαμάντσα που είναι από κάποιο εκδοτικό ίδρυμα εκεί, η Πιλάρ Μαρτίν είναι η καθηγήτριά τους και ήρθαν εδώ για να μας επισκεφτούν και για να μάθουν τι πάει να πει η Ευρώπη και τι έργο επιτελούμε εδώ εμείς που εκπροσωπούμε τον κόσμο και από πλευρά τη Εθνικών Κοινοβουλίων και από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ. Πέρα τη συνεδρία Καλό ταξίδι, καλό δρόμο.